Okay, everybody, in case you're wondering why I was waiting, it was because I know that we've got something that slipped off the agenda. Anyway. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. The adoption of the agenda. Πρώτο σημείο είναι η έγκριση της μερικής διάταξης. Με ενημέρωσα από το γραφείο της ηγητού Όλη Σμιτ ότι λόγω μιας διπλής ε, ακύρωσης ή καθυστέρησης πτήσης ε, δεν θα φτάσει η εγκαίρωση για την παρουσίαση της εκθεσής του που είναι στις 4 παρα 10, άρα το σημείο 6 της σημερινής ημερήσιας διάταξης θα αναβληθεί. Δεν μπορεί να γίνει η συζήτηση αργότερα σήμερα γιατί έχουμε τη δημόσια ακρόαση. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη, δεν βλέπω αντιρρήσεις, ωραία. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Ο πρώτος τριμερής ε, διάλογος για το ΕΜΙΡ έλαβε χώρα στις 10 Οκτωβρίου. Και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα, ιδίως ό,τι αφορά τη μεθοδολογία εργασίας και κάποια θέματα πολιτικά, τεχνικά και ούτω καθεξής. Επίσης καθορίσαμε τη διαδικασία, όπου είδαμε και εκεί κάποια τεχνικά σημεία και αυτά τα παραπέμψαμε σε μια ομάδα εργασίας η οποία θα μας δώσει τεχνικές πληροφορίες, τεχνικά στοιχεία πριν από τον επόμενο τριμερή διάλογο της 25ης Οκτωβρίου. Φυσικά δεν πρόκειται για λήψη αποφάσεων. Συγκρίνουμε και αντιπαραβάλλουμε προς το παρόν τα στοιχεία. Σημείο 3 της Μερισιάς Διάταξης, της έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέταση τροπολογιών. Θα δώσω το λόγο στον Αντρέα Σφάπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έκαναν τροπολογίες για την επικοδομητική τους εργασία. Είχαμε 67 τροπολογίες οι οποίες θα εμπλουτίσουν τη συζήτηση. Στην ε, ομάδα αυτή κρούσος για το ανταγωνιστικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξέρετε ότι προσπαθούμε να ε, μπορέσουμε μέσα μέσα στο χρόνο κάθε φορά να ε, εστιαζόμαστε σε ένα θέμα για να αποφύγουμε τις ε, γενικότητες και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Γι' αυτό και αποφάσισα εγώ στο σχέδιό μου να ε, παρουσιάσω ένα θέμα σχετικά με την οδηγία 1 του 2003 και να δούμε ε, πόσο μπορούμε όταν πρόκειται για αποζημιώσεις ε, να προχωρήσουμε εξοδικαστικά δικαστικά και πώς αποφασίζεται η χρηματική αποζημίωση και ποινή. Διότι ιδίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φοβάται ότι μία τέτοια εξοδικαστική λύση μπορεί να οδηγήσει σε μία κατάσταση όπου θα υπάρχει ένα παζάρι εκτός δικαστηρίου. Εγώ δεν έχω αυτή την πρόθεση όμως και αντιθέτως πιστεύω ότι ε, θα μπορέσει έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχυθεί στην προσπάθειά της και ε, να υπάρξει γρήγορα και αποτελεσματικά μία αποκατάσταση της ζημίας. Ε, δεν έχω ακούσει λοιπόν να υπάρχουν από αυτού του θέματος αντιρρήσεις και γι' αυτό ε, ίσως μπορεί να υπάρχει και μία τρίτη πτυχή όσον αφορά αυτές τις αποζημιώσεις και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν Ευχαριστώ προγράμματα ε, τα οποία ασχολούνται με τη διαδικασία συμμόρφωσης, compliance procedure, χωρίς όμως ε, να αποκλίνουν ε, από την επιτήρηση των καρτέλ. Επίσης το πρόγραμμα επίοικίες, leniency program πρέπει να μπορέσει εις το μέλλον να αντιμετωπίζεται πιο θετικά και ε, θα πρέπει να εφαρμόζονται και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά τρόπον ώστε ε, να μπορεί να επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση αρνήσεως, προξομήσεως αυτών των εγγράφων ε, το, ε, θα υπάρξει μια συζήτηση 8 Νοεμβρίου επί του θέματος και ε, όσοι ενδιαφέρονται ε, ευχαρίστως να συμμετάσχουν και επίσης θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο οποίος θα σχολιάσει επίσης και τέλος θα ήθελα εδώ να τοποθετηθώ στο θέμα ορισμένων ορισμένων τροπολογιών. Δηλαδή ε, πιστεύω ότι θα πρέπει οι τροπολογίες να έχουν συζητηθεί για να μπορέσουν να διεκπαιρεωθούν σωστά και αυτό όσον αφορά το collective redress, δηλαδή την ε, συλλογική επανόρθωση. Και το ίδιο θα ισχύει και για τις εναλλακτικές λύσεις των ε, διαφορών Alternative Dispute ε, Settlement και θα πρέπει ε, αυτές οι διαδικασίες να χρησιμοποιούνται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλά προτού επιβληθούν οι ποινές και κυρώσεις. Και ερχόμαστε έτσι στο επικουρικό δίκαιο και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα, μια κρατική ομπρέλα προστασίας ε, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται και γι' αυτού νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Υπάρχει και μια τροπολογία η οποία λέγει ότι όσον αφορά την, ε, ε, την ενέργεια και τις εταιρείες παραγωγής ενεργείας και των ε, οργανισμών πιστοληπτικής αξιολογήσεως είναι θέματα που θα πρέπει να εξετάσουμε και η Επιτροπή εδώ ανέφερε ότι θα πρέπει σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα θέματα αυτά. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι τα θέματα τα οποία δεν έχω ε, μέχρι στιγμής ε, θήξη. Ε, θα μπορέσουν να έχουν επίσης επιληθεί μέχρι την ψηφοφορία την οποία στην ημερομηνία δεν γνωρίζω ακόμη και είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο θέλετε. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τους άλλους εισηγητές, η Σόφη καταρχήν. Θα είμαι πολύ σύντομη. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτά που μας είπε ο εισηγητής. Συνεργαστήκαμε μια ομάδα δηλαδή εισηγητών και σκιωδών για την έκθεση για την ανταγωνιστικότητα και νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον ως προς τα βασικά ζητήματα Έριξα μια ματιά στις τροπολογίες και νομίζω ότι περισσότερες ε, είναι πολύ θετικές, ενισχύουν την έκθεση. Και στο θέμα των συλλογικών αγωγών θα ήθελα να πω ότι φτάσαμε σε πολύ καλούς συμβιβασμούς και ως προς υπηρεσίες και υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος ίσως υπάρχουν περισσότερες διαφωνίες διότι δεν είμαστε υπέρ των ε, ΔΕΚΟ και δεν θέλουμε να νομοθετήσουμε, δεν θέλουμε ένα πλαίσιο, αλλά σε αυτό πάντα διαφωνούσαμε και έτσι θα συνεχίσουμε. Στο θέμα της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω υποβάλει μια σειρά τροπολογιών τις αναφέρατε χωρίς να πείτε αν τις υποστηρίζετε ή όχι. Πρόκειται για μια προσπάθεια για να έχουμε προτάσεις που να δίνουν καλύτερη διάρθρωση στη συνεργασία, διότι κάθε χρόνο εγκρίνουμε την έκθεση ανταγωνισμού και άλλες συναφείς εκθέσεις και η Επιτροπή μας λέει ευχαριστώ, ευγενέστατα και μετά κάνει αυτό που θέλει στο 99% των περιπτώσεων υποστηρίζω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν υπάρχει δημοκρατική εποπτεία, ουσιώδης δημοκρατική εποπτεία και αν δείτε την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας και την τροπή που παίρνουν οι συζητήσεις για περισσότερη οικονομική ολοκλήρωση και συντονισμό, Βλέπουμε ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο input, περισσότερα δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορώ να δεχτώ ε, και άλλες προτάσεις, αλλά αυτή ήταν η δική μου συνεισφορά. Ντέρκ, θέλεις το λόγο? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σφάμπ για το προσχέδιο έκθεσης και όπως είπα και πριν υποστηρίζω τα περισσότερα τμήματα του σχεδίου και θα αναφερθώ στις δικές μας τροπολογίες. Στην ετήσια έκθεση περί ανταγωνισμού 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρθηκε στις ανησυχίες ως προς τα προσωρινά μέτρα που μπορεί να μην είναι και τόσο προσωρινά. Επίσης τονίσαμε την ανάγκη να αρθούν οι εξαιρέσεις το ταχύτερο δυνατό αλλά είδαμε ότι είχαμε μία περαιτέρω παράταση κρατικών ενισχύσεων και στις 6, 12 και 14 το τονίζω αυτό. Στα αντιτράστ πιστεύω ότι η πολιτική κυρώσεων της Επιτροπής θα πρέπει να βελτιωθεί και θα πρέπει να έχουμε και άλλα μέσα κυρώσεων πέρα από τα χρηματικά ποσά. Και δεν θα πρέπει να βασίζεται η Επιτροπή σε θέματα ανταγωνισμού χωρίς να λαμβάνει υπόψη οι οικονομικές ε, επιπλοκές. Οι, Γκρέσλε και Ρεβελίνη έχουν δύο εκθέσεις που θα ψηφιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η τροπολογία 44 μιλά για την εφαρμογή των κυρώσεων και στον τομέα του προϋπολογισμού. Αυτό όμως οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων και άρα αμφισβητούμε την αμεροληψία της Επιτροπής, διότι κινείται πέρα της εντολής του ανταγωνισμού. Ως προς την τροπολογία μου 37, αν υπερψηφιστεί, θα θεωρήσουμε ότι οι κυρώσεις δεν είναι εναλλακτικός μηχανισμός. Ελπίζω το πνεύμα αυτών των σημείων να ενταχθεί στην τελική έκδοση της έκθεσης περί ανταγωνισμού και ως προς τις συλλογικές προσφυγές την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση ο εισηγητής ήταν συνεργάσιμος και έτσι φτάσαμε σε ικανοποιητικές λύσεις ως προς τα περισσότερα ζητήματα και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ε, διότι ήταν ανοιχτός σε πολλές υποδείξεις. Φίλιπ Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντρέα για την πολύ καλή έκθεσή του. Συμφωνώ και εγώ με την ιδέα να μην έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα ευχολόγιο στην έκθεση ανταγωνισμού. Το έχουμε κάνει και κατά το παρελθόν αυτό. Α εστιάσουμε λοιπόν περισσότερο σε ορισμένα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε τη ουσία στα πρόστιμα. Ε, βλέποντας ε, το σημερινό πλαίσιο, βλέπουμε ότι η εστίαση τελικά ήταν ε, στα μέτρα τα οποία ελήφθησαν για τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Εμένα αυτό με ανησυχεί περισσότερο αν δω τον ε, μάκρο αντίκτυπο στην ε, πολιτική ανταγωνισμού. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο αντίκτυπο όλων αυτών των κρατικών ενισχύσεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα είναι ένα πολύ πιο μείζον θέμα από αυτό των προστήμων. Άρα βλέπετε ότι είναι διαφορετική η εστίαση ανάλογα με τις προτεραιότητες που έχει ο καθένας μας. Ελπίζω όμως να καταλήξουμε ε, σε μια καλή έκθεση. Για τη Σοφή τώρα, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, είπες ότι είσαι αντίθετη στο να υπάρχει μια οδηγία πλαίσιο για τις υπηρεσίε γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Για μια φορά ε, είμαστε σε αντίθετα στρατόπεδα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιούργεν θέλω το λόγο για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Άργησα λιγάκι, αλλά νομίζω ότι συζητάμε την έκθεση ανταγωνιστικότητος. Σαν μικρή ομάδα πολλές φορές ε, είμαστε πολύ πιεσμένοι από πλευράς εργασίας και γι' αυτό δεν προλάβαμε να διατυπώσουμε τροπολογίες. Κοίταξα όμως τις τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα και το σχόλιο μου είναι ότι αυτά που είπε ο Φιλίπ Λομπέρ σχετικά με τις ενισχύσεις, ιδίως εάν δίδονται σε τράπεζες θα πρέπει να στηρίζονται με πολύ σαφή έγγραφα και θα πρέπει να υπάρχει υπάρχει παρακολούθηση και ένα δεύτερο θέμα επ' αυτού είναι ότι ε, όσον αφορά την παροχή ενεργείας ε, έχει γίνει μία τροπολογία την οποία ε, και εμείς στηρίζουμε σχετικά με την ε, την αποφυγή ολιγοπολίων ε, αυτές είναι προτάσεις οι οποίες από την πλευρά μας είναι ε, άξιες να στηριχθούν και περισσότερα δεν έχω να σας πω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ η Άντελιν. Ο Άντελιν, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι ο αρμόδιος Θα ήθελα εγώ να αναφερθώ στην τροπολογία τη δική μου και ε, καταρχάς να μιλήσω για τις συλλογικέ προσφυγές, ένα ζήτημα από το οποίο συνεδριάσαμε, η ομάδα εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασε και καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία επί της ουσίας και σίγουρα η συμφωνία αυτή ε, θα αντικατοπρίστε φαντάζομαι και στην παρούσα έκθεση. Άρα νομίζω ότι πηγαίνουμε προς μία ε, συμβιβαστική λύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, φυσικά και θα πρέπει να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα. Επομένως, στο βαθμό που τα πρόστιμα δεν έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα, ε, πρέπει να δούμε τι κίνητρα, πώς αποτελούν κίνητρο. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Επίσης, οι διαδικασίες συγκέντρωσης ε, θα πρέπει να διέπονται από τη λογική της ε, αγοράς. Η Λίσα Φερέιρα έχει κάνει κάποια σχόλια που δεν είναι παρούσα εδώ πράγματι να μην είναι χριστιανιάτικο δέντρο κάθε χρόνο η έκθεση αυτή, αλλά πρέπει να εντοπίσονται τα βασικά ζητήματα και να υπάρχει μια συνέχεια. Ε, αυτά λοιπόν λέει η Λίζα Φερέιρα ε, σε ό,τι αφορά ε, τα προηγούμενα ζητήματα, σε ό,τι αφορά και τους οίκους αξιολόγησης και σε ό,τι αφορά την κατάρχηση δεσπόζουσας θέσης. Είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα, ιδίως για το γεωργοδιατροφικό τομέα. Και η Λίζα Φερέιρα έχει κάνει και μια άλλη τροπολογία για την τραπεζική κρίση και την ε, λύση που ε, προτείνει και η οποία νομίζω ότι είναι εύστοχη και θα πρέπει να τη λάβει υπόψη ε, ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Τόμας Μάν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συγχαίρω τον Ανδρέα, ο οποίος κατάφερε με τους σκιώδεις να καταλήξει σε σύμπνοια. Ε, σύμφωνο και αν πρόκειται για αποζημιώσεις και για κυρώσεις θα πρέπει να έχουν μία αποτρεπτική ε, λειτουργία και δεν θα είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει κανείς να θεωρεί ότι θα ξεμπλέξει εύκολα. Υπάρχουν διαδικασίες και βλέπω ότι έχετε συμφωνήσει ε, και όσον αφορά τις τροπολογίες επίσης ε, ε, συμφωνώ αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ καταρχήν στις rating agencies, στις εταιρείες χρηματοληπτικής, αξιολογήσεως χρηματοληπτικής ικανότητας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτές πρέπει να περιληφθούν εδώ στον ανταγωνισμό διότι έχει παρανοηθεί η δημιουργία ενός τέτοιου ευρωπαϊκού γραφείου διότι εάν το γραφείο αυτό καταρτιστεί και εξαρτάται από πολιτικές αποφάσεις και δεν αποδίδει στον στόχο που θέλουμε εμείς, καλύτερα είναι να το ξεχάσουμε διότι βλέπουμε εδώ ότι σε αυτές τις rating agencies συμμετέχουν και εκατομμυριούχοι, καταλήγουν σε αποφάσεις που μας καταπλήσουν. Ε, υπάρχουν βέβαια και άλλες μικρότερες τέτοιες, μικρότερες τέτοιες ε, εταιρείες και πιστεύω ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ευρωπαϊκό όργανο πολιτικής παρεμβάσεως διότι δεν θα είναι προς όφελός μας. Έχω μιλήσει επίσης ε, με ορισμένους σχετικά με τις ασφάλειες που μας λένε ότι πρόκειται για γίγαντε αλλά οι ασφαλιστικές αυτές εταιρείες πρέπει να ακολουθούν τις αποφάσεις των rating agencies. Δεν έχουν ε, δυνατότητα ελιγμού και δεν είναι ε, δυνατόν να τους επιβάλλονται οι πολιτικές των καταθέσεων και τοποθετήσεών τους. Ε, και πολύ σωστά ο Ανδρέας είπε διάφορα αλλά στην τροπολογία 16 είπε να υπάρχει ένα ταμείο με ε, ίδια χρηματοδότηση για την εξυγίαση των επιχειρήσεων που απειλούνται από ε, χρεοκοπία. Θα ήθελα να ξέρω τι μορφή θα έχει αυτό. Αν κάποιος έχει χρεοκοπήσει έχει καλός αλλά εάν απειλείται με χρεοκοπία τι θα γίνει, θα παρεμβαίνει κανείς στην αγορά. Έχω ένα μεγάλο ερώτηματικό και είναι κάτι που θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε. Και τέλος θα καταλήξω με τις παρατηρήσεις που κάνω και σε άλλες επιτροπείς. Είναι μία έκθεση κατά πρωτοβουλία, συζητιέται τις Δευτέρες όπου υπάρχουν ελάχιστοι εκεί. Μπορούμε να την διαγράψουμε και να καταστηθεί μία σωστή έκθεση η οποία θα εξεταστεί στο Στρασβούργο σοβαρά στον κατάλληλο χρόνο και και ε, δεν είναι μια διαδικασία που αξίζει να χρησιμοποιηθεί σαν να είναι catch the eye. Λοιπόν, Ανδρέα είσαι έξυπνος, είμαι σίγουρος ότι θα βρεις κάποια καλύτερη λύση. Ανδρέα έχεις εσύ το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήρθε και ο Γιώργος, τον οποίο δεν τον είχα δει. Θα είμαι πολύ ε, σύντομος για να ακούσουμε τον ε, Ανδρέας, γιατί θα ήθελα να τον συγχαρώ για την εξαιρετική αυτή εργασία. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι μείζονο ε, σημασίας. Θα ήθελα να αναφερθώ στις τροπολογίες μου που αφορούν τον τομέα του διαδικτύου γιατί ακόμα και σε μία τέτοια έκθεση γενικής εμβέλειας θα πρέπει να αναφερθούμε σε επιμέρους τομείς. Και θα ήθελα να επισύρω την προσοχή στα ολιγοπόλια στις αγορές, διότι κάνουν καταχρήσεις, δεν προβάλλουν καινοτομίες, δεν παρέχουν σωστές υπηρεσίες και ζημιώνουν τους καταναλωτές και τις αγορές. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες αντιμετώπισης αυτών των ολιγοπολίων. Και εδώ αναφέρομαι και στους οίκους πιστοληπτικής ικανότητας. Γι' αυτό θα ήθελα να λάβετε υπόψη την τροπολογία για τα ολιγοπόλια και να την μεταχειριστεί ανάλογα και ο εισηγητής μας. Τώρα έχει το λόγο Ανδρέας. Ευχαριστώ. Βεβαίως όλες οι τροπολογίες θα εξεταστούν πάρα πολύ προσεκτικά ε, και πέραν αυτού όμως πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο να το περικόψουμε, να το έχουμε πιο εστιασμένο από ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν και από αυτού συμφωνούμε όλοι. Δεν έχει, καμία, δεν έχει κανένα νόημα ε, κάθε χρόνο να κάνουμε μία έκθεση η οποία καταλήγει ε, στον κάλαθο των αρχίστρων και θα πρέπει να σε λίγα πράγματα συγκεκριμένα. Φιλίπ, σχετικά με την, ε, τις κυρώσεις κατά τον καρτέλ το έχουμε συζητήσει διότι πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για τον ανταγωνισμό ε, αλλά θα πρέπει να περιληφθούν και άλλοι τομείς ε, εγώ όμως θα ήθελα να εστιαστώ εδώ σε δύο-τρεις και να μην πλατιάσω μετά αυτό που είπε ο συνάδελφος Πλασέντο έχει δίκιο. Θα πρέπει να υπάρχει ε, μία αποτρεπτική λειτουργία των κυρώσεων ε, και των προστήμων αλλά ε, οι ζημιωμένοι τελικά βγαίνουν χαμένοι και γι' αυτό θα ήθελα να ελέγξουμε την πρόταση και να δούμε σε περίπτωση μιας εξοδικαστικής διευθετήσεως αν μπορεί να υπάρξει ένα έλεγχος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλά πρώτης εποβολής του προστήμου για να μπορεί κανείς να καταλήξει σε μια δίκαιη λύση και να μην κλείνει η πλάστιγκα υπέρ των καρτέλ. Σε άλλα θέματα δεν χρειάζεται ίσως να σχολιάσω τώρα όταν οι συνάδελφοι που έθεσαν τις ερωτήσεις έχουν φύγει αλλά πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αποτελεσματικά βάσει των συνθήκων ΕΟΚ ε, και κύριε Λάμπερτς βέβαια η μελέτη την οποία ζήτησε το Κοινοβούλιο δεν απέδωσε ε, αυτά τα οποία εμείς αναμέναμε και δεν μπορεί να μας καθοδηγήσει ε, σχετικά με το δίκαιο των ενισχύσεων προς τις τράπεζες και χρειαζόμαστε ε, από εκεί ε, κάτι παραπάνω για να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω όμως ότι μέχρι τις τέσσερις εβδομάδες που θα περάσουν ώσπου να γίνει η ψηφοφορία κάπου θα έχουμε καταλήξει σε εμβαστικές τροπολογίες. Λέγεται ότι θα ψηφίσουμε, λέει πρόεδρος, 22 Νοεμβρίου για να έρθει στην ε, Ολομέλεια του Δεκεμβρίου και τώρα έχουμε να ψηφίσουμε. Θα σας δώσω λίγο λίγα λεπτά για να βρείτε τις κάρτες σας στις ψηφοφορίες και να τις τοποθετήσετε στη θέση τους. Το λοιπόν, πρώτο θέμα είναι η μεταρρύθμιση των κανόνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι κρατικέ ενισχύσει, τι υπηρεσίε γενικού οικονομικού συμφέροντο. Οι κάρτε είναι όλε στη θέση του. Λοιπόν, έχω ξεμείνει λίγο μόνο μου εδώ. Λοιπόν, για να δούμε πώς μπορούμε. Ο Άντολιν δεν έχει κάρτα. Μείον ένας λοιπόν, ως προς τις κάρτες. Can Λοιπόν, δοκιμαστική ψηφοφορία. Σας παρακαλώ, πατήστε το κουμπί. Ούτε εσείς έχετε την κάρτα σας. Yes, Sophie, fine. Oui. Ακούστε, σε ό,τι αφορά την ε, ψηφοφορία της εκθέσεως του Πίτερ Σάιμον, δεν αναφέρεται στις οδηγίες, αλλά το ΕΛΚ στηρίζει όλες τις συμβιβαστικέ. Yes. Ashley, κάτι και εσύ μου κάνεις κάποιο νόημα. Ναι, έχω ξεχάσει την ε, κάρτα μου και όταν ε, είναι λίγο αμφίροπο το αποτέλεσμα θα σηκώνω το χέρι μου, αν Λοιπόν, ωραία. Έχουμε λοιπόν δύο συναδέλφους χωρίς κάρτα, Ashley και Άντολιν. Κάποιος άλλος. Γιούργεν. Jürgen also hasn't got his. Και ο Jürgen. Αμφίρω από το αποτέλεσμα θα πρέπει να ξαναψηφίζουμε ή να δεχόμαστε τις ξεχωριστές αυτές ψήφους διανατάσεως χειρός. Λοιπόν, 31 ε, έχουν ε, εισάγει τις κάρτες, δεν ψήφισαν όλοι όμως. Okay. Anyway, we'll start. Τέλος πάνω, θα ξεκινήσουμε παρόλα αυτά. Παράγραφος 1. Τροπολογία 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Νομίζω. Ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Η Άλντε έχει έναν παραπάνω. Άρα δεν θα ψηφίζω εγώ. Αν και θα ανεπέμενα θα μπορούσα και να ψηφίσω τέλος πάντων. Λοιπόν, πέραση ψηφοφορία. 19 ψήφοι υπέρ 10 κατά. Άρα και οι τρεις που δεν έχουν κάρτα δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα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 61 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. Συμβαστική Β, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές,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 εγκρίνεται. Πού είναι η συμβαστική δέλτα, μπι λατινικό. Μάλιστα, τη βρήκα. Επιτέλους, μετά από πολλές σελίδες. Λοιπόν, συμβαστική δέλτα, D, ψήφι περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 38, υπέρ, κατά, αποχές, Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Τροπολογία 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα πρέπει να το ελέγξουμε. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Οι μεσαίοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Ναι, συγγνώμη που δεν σας ανακοίνωσα λίγο. Το αποτέλεσμα ήταν 20 υπέρ, 11 κατά. Νόμιζα ότι φαινόταν στην οθόνη. Λοιπόν, τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ, κατά, αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε την τροπολογία 41, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 20 υπέρ, 12 κατά είναι το αποτέλεσμα. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Μα δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Πω, δεν θα γίνει έτσι. Τέλος πάντων κάποιοι σηκώνουν, αλλά όχι αρκετοί. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. 20 ψήφοι υπέρ, 11 κατά. Άρα, όταν δεν σηκώνετε τα χέρια σας, να υπολογίζω 20 ψήφους υπέρ. Λοιπόν, πέμπτη ε, συμβαστική ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 49, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεν κατάλαβα το αποτέλεσμα, το ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. 17 ψήφοι υπέρ, 15 κατά. Λείπει κάποια κάρτα. Άρα 17 υπέρ, 16 κατά με τον Άσλι. Για μισό λεπτό. Right. We've got... Don't press the button yet. It's, it's 17... Λοιπόν, 17 είχαμε υπέρ, 15 κατά. Τώρα, ποιοι άλλοι είναι υπέρ που δεν είχαν κάρτα. Άντολιν, Πίτερ, είστε κατά. Άρα έχουμε άλλους τρεις που είναι αντίθετοι. Ο Γιούργεν κατά. Απορρίπτεται επομένω. Απορρίπτεται. Με 19 ψήφους κατά. Αυτό ήταν το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε. Τροπολογία 6. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική σιγματά λατινικο F, τμήμα. Τα Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G, Z, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H, λατινικό ή Πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 71 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 16 ψήφοι υπέρ, 17 κατά. Άρα δεν γίνεται δεκτή. Ήμκο 9 τροπολογία υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 7 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική α, λατινικό θήτα ελληνικό. Υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 82 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, από συμβιβαστική J για το ελληνικό υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο παραγράφου 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω όλα στο ελέγξουμε καλύτερα. 113. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 17 υπέρ, 17 κατά. Έξτρα έχουμε κάποιον. Άλλον ένα κατά. Ούτως ή άλλως Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 115. Παρακαλώ. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Σας είχαμε υποβάλει και προηγουμένως την τροπολογία 15 ε, και θα ήθελα εδώ να προσθέσω με προφορική τροπολογία ε, ε, επιδοτήσεις αντισταθμιστικές και ε, να υπάρχει μία ανταλλαγή με τις επιχειρήσεις. Είναι ε, μία προφορική τροπολογία η οποία ε, έχει συζητηθεί και με το ΕΛΚ. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν μιλάμε πλέον για επιδοτήσεις και νομίζω ότι αλλάζοντας την ορολογία θα μπορέσουμε όλοι να συνενέσουμε σε αυτή την τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις στην τροπολογία αυτή. Άρα την ψηφίζουμε. Έχετε καταλάβει πριν μας πρόκειται όλοι. Λοιπόν, προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. αντί τις 115. Τι θέλετε, να ψηφίσουμε και την 115. Γιατί, δεν κατάλαβα. Yes. The, yeah, the oral amendment. Η προφορική τροπολογία που μόλις ψηφίσαμε αντικαθιστά την τροπολογία 115 γιατί κανείς δεν ήταν αντίθετος σε αυτό. Ναι, αλλά εδώ ε, είπε ότι συμφωνήθηκε σαν αντικατάσταση ενώ εμείς θέλουμε να ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία που ανέφερε ο συνάδελφος Ζήμων. Καλώς. Άρα τι ψηφίσαμε την προφορική τροπολογία που μόλις υπέβαλε ο κύριος Σίμων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 Α, έχουμε και άλλο τμήμα. Έκτο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπάρχει και έβδομο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι υπέρ όλων αυτών των ε, χωριστών τμήματων ε, των συμβιβαστικών. Δεν θα το δεχθώ στο μέλλον και σημειώστε το παρακαλώ. Για να πάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Επί 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Την τροπολογία 6. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. 21 ψήφοι υπέρ, 15 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο στις ιδεολογικές αναφορές 1-12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται αρχικό κείμενο 13-15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. 27 ψηφί υπέρ, 8 κατά, μία αποχή. So congratulations to Πρόεδρε, πολύ ε, γρήγορα. Είπατε ότι δεν θα επιτρέψετε πλέον split vote. Θα το εφαρμόσετε τώρα γιατί η πολιτική σας ομάδα έχει ζητήσει ένα τέτοιο split vote. Εγώ ευχαρίστως να το εφαρμόσουμε αμέσως. Λέω ότι στο μέλλον, στο μέλλον την επόμενη φορά που θα ψηφίσουμε δεν πρέπει να έχουμε τόσες ξεχωριστές ψηφοφορίες στα, στις τροπολογίες συμβασμού. Αυτό αναφέρεται στον κανονισμό και όταν υπάρχει διαχωρισμός σε 5, 6, 7 τμήματα, εάν το είχα δει εκ των θα το είχα αποκλείσει. Αλλά τώρα δεν μπορώ να το κάνω στο μέσον της ψηφοφορίας. Δεν μου επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Ε? Um, I'm going to Λοιπόν, η ΑΛΔΕ υποστηρίζει τροπολογία στην ΑΒ, β, c, d, e, h και i. Η φιλελεύθερη, κάτι το οποίο δεν φαίνεται στο κείμενο και το οποίο θα προσθεθεί. Ψηφίζουμε τώρα προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της συλλογικής προσφυγής. Ε, τροπολογία α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ο συμβιβασμός. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβασμού Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού D σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία συμβασμού ε, υπέρ, ε υπέρ, κατά, κάποιοι φαίνεστε χαμένοι. Είμαστε στην τροπολογία συμβασμού ε. Ε, λοιπόν. Την ψηφίσαμε την ε, Δέλτα σε δύο τμήματα. Ψηφίσαμε σε δύο τμήματα. Το πρώτο εγκρίθηκε, το δεύτερο απορρίφθηκε. Τώρα βρισκόμαστε στην ε Ποιος θέλει το λόγο? But we got some Φαίνεται, Αντολίν, εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια σύγχυση. Αντολίν. Στο Δέλτα, στο δεύτερο τμήμα, θα πρέπει να ξαναγίνει η ψηφοφορία. Στο Δέλτα, στο δεύτερο, θα πρέπει να ξαναγεί. Ναι, στο Δέλτα, Δέλτα εννοούσα. Στο Δέλτα θα πρέπει να ξαναγίνει ψηφοφορία διότι στο δεύτερο τμήμα ε, οι περισσότερες ομάδες ε, έχουν ταχθεί υπέρ και φάνηκε αρνητική η ψήφος. Νομίζω ότι θα πρέπει να επαναληφθεί λοιπόν γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Θα ελέγξουμε λοιπόν, θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα λοιπόν της ΔΕΛΤΑ. Δεύτερο τμήμα της ΔΕΛΤΑ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 27 υπέρ 8 κατά. Πράγματι έχει εγκριθεί. Τώρα είμαστε στην ε, υπέρ της ε, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θα ελέγξω, θα ελέγξω αν το επιθυμείτε. 17 ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 20 υπέρ, 15 κατά. Συμβασμός F, σίγμα τάφσε τρία τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ του πρώτου, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ της 25 κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε γιατί δεν είμαι και σίγουρη. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 16 υπέρ, 18 κατά και μία αποχή. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάποιον που έχει πρόβλημα με την κάρτα του. Απορρίπτεται λοιπόν. Ναι, 16-18 το είπαμε. Άρα απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές απορρίπτεται. Ωραία, αν θέλετε ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίστε όσο τρέχει. 18 υπέρ, 16 κατά. Μία αποχή. Άρα εγκρίνεται. Συμβιβασμός Ι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 33 υπέρ. Μία ψήφος κατά και καθόλου αποχές. Σας ευχαριστώ. Και να συγχαρούμε τον εισηγητή. Όπως είπα και νωρίτερα, το 6 δεν θα συζητηθεί η ετήσια έκθεση για τους φόρους. Μετατίθεται. Άρα θα διακόψουμε μέχρι τις 4.30, οπότε και θα αρχίσει η δημόσια ακρόαση για την οικονομική διακυβέρνηση. Λοιπόν, μισή ώρα διάλειμμα. Καλησπέρα σας. Άφησα λίγα ακόμη λεφτά να περάσουν διότι ήθελα να δω αν θα έφταναν κι άλλοι ευρωβουλευτές αλλά τώρα έχουμε μία ακρόαση σχετικά με τη διαχείριση κρίσεως και την οικονομική διακυβέρνηση. Δηλαδή έχουμε δύο συνεδρίες, μία ομάδα που θα συζητήσει για τη διαχείριση κρίσεως ε, τον Αντρέ Σαπίρ και τον Ρικάρντο Καμπράλ 10 λεπτά εκαστός και μετά ερωταπαντήσεις και μετά από μία ώρα θα προχωρήσουμε στη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα με τον Γιούργεν Στάρκ και τον Ζερόμ Κρίλ οι οποίοι είπαν ότι ευχαρίστως να ακούσουν και το πρώτο, την πρώτη στρογγυλή τράπεζα γιατί τους ενδιαφέρει και ενδέχεται να έχουν να μας κάνουν πολύ πιο εμπεριστατωμένα σχόλια οπότε ευχαρίστως θα τους δώσω το λόγο. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση αλλά προσπαθούμε να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα μαζί που είναι δύσκολα τα πράγματα και προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε και όλες τις πληροφορίες Γι' αυτό και αποδίδουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία σε ορισμένα πράγματα από ό,τι νομίζετε. Ευχαριστώ λοιπόν τους ομιλητές και ε, ε, το ρολόι ε, μετράει το χρόνο σας και όταν μηδενιστεί σημαίνει ότι έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Ο Ντρέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να έρθω στην Επιτροπή σας. Τρία ερωτήματα μας ετέθησαν σχετικά με τη διαχείριση κρίσεως. Η πρώτη αναφέρεται στον κίνδυνο διπλής υφέσεως και το τι μπορούμε να κάνουμε double deep ε, recession και μετά τι μελγενέστε με την ε, ε, Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία και θα προσπαθήσω να ασχοληθώ με όλα αυτά τα θέματα και ιδίως περισσότερο με τις τέσσερις χώρες στην αρχή διαβάζω στην ε, ε, έκθεση του 2003 ε, μία σύντομη παράγραφο σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμενο ότι σχετικά με ε, τον δημοσιονομικό συντονισμό λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ετοιμάζει προγράμματα ε, εθνικής σταθερότητος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και των κρατών μελών και της Ευρωζώνης και άπειρας και καταρτιστούν αυτά τα προγράμματα μπορούν να παγιωθούν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σταθερότητος που μπορεί να ε, καθορίσει την φορολογική πολιτική και ε, μία τέτοια διαδικασία θα διευκολυνθεί με το να ε, διαιρέσουμε στους 12 μήνες του ευρωπαϊκό εξάμεινο και να υπάρχει ένα εθνικό εξάμεινο όπου θα παρεμβαίνουν οι παράγοντες που αναφέρονται σε την εθνική πολιτική. Τώρα έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά θα έρθουμε έτσι στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, δηλαδή ότι ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής σταθερότητας, δεν έχουμε φτάσει δηλαδή στο σημείο όπου εάν συνδυάσουμε τα εθνικά προγράμματα και δούμε τι σημασία έχουν για τον, ε, την Ευρωζώνη στο σύνολό της, μπορούμε στη συνέχεια να ε, ε, μπορούν στη συνέχεια τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτές τις προβολές για να καταρτήσουν τον εθνικό προπολογισμό. Άρα μία έννοια ενός πολιτικού μείγματος που αποτελεί από διάφορα τμήματα από κάτω προς τα πάνω και όχι αντιστρόφως ένα τέτοιο πολιτικό μείγμα μπορεί να είναι χρήσιμο και θα μπορέσει να επιλύσει διάφορα προβλήματα. Ε, βέβαια πρέπει να πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και το ευρωπαϊκό εξάμεινο μπορεί να επηρεάσει να αποφύγουμε την διπλή ύφεση ε, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε καταφέρει. Άρα, ε, ποια είναι η κατάσταση στις χώρες όπου υπάρχει ένα πρόγραμμα. Θα προσπαθήσω να τονίσω ε, προς ε, τα μέλη της Επιτροπής την διάκριση μεταξύ της Ελλάδος από τη μία πλευρά και των δύο άλλων χωρών που είναι στο πρόγραμμα της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Εάν εξετάσω την Ελλάδα για λόγους οποίους θα παρουσιάσω στη συνέχεια ήταν σαφές από την αρχή ότι αυτό όπως μου είπε κάποιος αυτό θα είναι ένας μαραθώνιος δηλαδή θα χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος για να μπορέσει και η ευρωπαϊκή πλευρά και η ελληνική πλευρά και ιδίω αυτή η δεύτερη να ε, διατυπώσει τις μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να αντεπεξέλθει της κρίσεως και να μεταρρυθμιστεί. Θα ήταν ε, λοιπόν όντως ένας μαραθώνιος, αλλά υπάρχει μία αντίφαση, διότι η διαδικασία έχει τοποθετήσει διάφορα ορόσημα τα οποία είναι πολύ βραχυπρόθεσμα και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι κάθε τρίμηνο αναρωτιόμαστε αν η Ελλάδα θα καταφέρει να επιτύχει το ορόσημο που έχει τεθεί. Εάν έχετε έναν μαραθώνιο δεν ε, κοιτάτε σε κάθε τέταρτο μιλίου ε, εάν είσαστε στο χρόνο σας. Ε, πρέπει να είναι πιο μακροπρόθεσμη η προοπτική και από ευρωπαϊκής πλευράς και από ελληνικής πλευράς για να υπάρχει ο χρόνος να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Ε, επίσης δεν χρειάζεται να σας παρακολουθεί η αγορά κάθε τέταρτο μιλίου για να δει αν επιτυγχάνετε τους στόχους και στην αρχή ε, ε είχε λεχθεί ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να επιστρέψει αγορές το 2012. Ήταν λανθασμένη αυτή η εκτίμηση. Επιτρέπεστε μου λοιπόν να σας πω γιατί η Ελλάδα θα παραμείνει ε, στον μαραθώνιο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να μεταρρυθμιστεί αλλά αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα δεν υπάρχει ικανοποιητική διοίκηση και η ε, World Bank, η ε, Παγκόσμια Τράπεζα έχει δημοσιεύσει έναν δείκτη για τις επιχειρήσεις που αξιολογεί τη διοικητική κατάσταση στις διάφορες χώρες. Από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης η Ελλάδα έχει τη χειρότερη βαθμολογία με έναν δείκτη 56 είναι ο αριθμός τον οποίο έχουν επίσης η Αλβανία και η Λευκορωσία και αυτή είναι η βαθμολόγηση της Παγκοσμίου Τραπέζης για την Ελλάδα. Αν δείτε την επόμενη χώρα της Ευρωζώνης, η Πορτογαλία είναι στο 70, δηλαδή είναι αρκετά πιο προηγμένη από την Ελλάδα σε αυτό το τομέα. Εάν κοιτάξετε έναν άλλο δείκτη, την οικονομική δομή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν κοιτάξτε τη συμμετοχή της απασχόλησης σε εταιρείες με λιγότερο των 10 εργαζομένων αν μιλάμε για τη Γερμανία λέμε ότι η Γερμανία έχει πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά αυτές δεν είναι πολύ μικρές δηλαδή κάτω των 10 απασχολουμένων το 90% στην Ελλάδα είναι κάτω από 10 ε, απασχολουμένους το 58% για την ακρίβεια της απασχόλησης στην Ελλάδα είναι σε μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων και καταλαβαίνετε έτσι ποια είναι η δομή παραγωγής. Η Πορτογαλία η οποία ε, ε, ε, είναι στο 41% βλέπετε ότι υπάρχει με ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ της Ελλάδος και της Πορτογαλίας και όταν μιλάμε για το άνοιγμα προς τα έξω της οικονομίας για τα αγαθά και υπηρεσίες σε σχέση με το ΑΕΠ βλέπουμε επίσης ότι όλες οι οικονομίες η Ιρλανδία και άλλες έχουν ένα πόσο ποσοστό εξαγωγών περίπου στο 80% σε σχέση με το ΑΕΠ. Και μετά έχετε την Ελλάδα η οποία πάλι έχει τη χειρότερη βαθμολόγηση και το χαμηλότερο ποσοστό των χωρών της Ευρωζώνης ακόμη και των μικρών. Δεν είναι δηλαδή μια μικρή ανοιχτή οικονομία, είναι μια μικρή κλειστή οικονομία. Μόνο 20% σε σχέση με το 23% ε, ε, είναι ε, προς τα έξω σε εξαγωγές. Χρειάζεται λοιπόν μία μεταρρύθμιση τεράστια της οικονομίας η οποία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια και το πρόγραμμα που καταρτίστηκε στην αρχή δεν ήταν λογικό. Δεν σας λέω ότι δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί. Βεβαίως μπορεί να μεταρρυθμιστεί και όλα τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αναμορφωθεί αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Όταν λοιπόν λοιπόν κοιτάμε την πρόοδο, το πρόγραμμα και βάζουμε την Ελλάδα σε μια τελείως διαφορετική κατηγορία από τις άλλες δύο χώρες, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, είναι σε μια δυσχερή θέση και θα χρειαστεί χρόνο. Δεν θα υπάρχει ένα γρήγορο ξεμπέρδεμα, γιατί όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο θα έχει δυσάρεστες εκπλήξεις και αυτό το βλέπουμε κάθε εβδομάδα. Όταν βλέπουμε ότι η Ελλάδα όλο και ε, ε, διολυσθένει διότι οι αρχικές ε, προσμονές δεν ήταν λογικές οι αρχικές προσδοκίες. Μας είπατε να μιλήσουμε και για το EFSF και το ESM που είναι ο διάδοχός του σαν σύστημα. Θα μπορούσα να πω και πάλι για αυτά που είπα για την Ελλάδα ότι η Ελλάδα από την αρχή επρόκειτο να οδηγηθεί στη χρεοκοπία και ήταν λογικό να εφαρμοστούν τα προγράμματα τα οποία εφαρμόστηκαν. Δεν θα θίξω το θέμα αυτό, δεν θέλω να το συζητήσω παρόλο που αξίζει να το προσέξουμε. Αλλά η κατάσταση της Ελλάδος είναι τελείως διαφορετική από από τις άλλες δύο χώρες που είναι στο πρόγραμμα, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας και βεβαίως από την κατάσταση της Ιταλίας παραδείγματος χάρη και της Ισπανίας. Εξού και όταν εξετάζουμε το ρόλο του EFSF και του ESM στο μέλλον θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση διότι εγώ είμαι βέβαιος ότι το θέμα αυτό θα ανακύψει και στη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα. Ε, ε, έχω την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να διαδραματίσει έναν κρίσιμο ρόλο μαζί με τις φορολογικές αρχές. Δηλαδή έχουμε το ρόλο της ΕΚΤ ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και ήδη από, για όλη την περίοδο από το 1999 δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το ρόλο της ΕΚΤ σε φυσιολογική εποχή με το ρόλο μιας κεντρικής τράπεζας σε περίοδο κρίσεως διότι το σύστημα αυτό δεν είχε επινοηθεί για καταστάσεις κρίσεως όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά κανένα από αυτά τα συστήματα γι' αυτό και συνέχεια πρέπει να συζητήσουμε στη διακυβέρνηση πώς θα λειτουργήσουμε σε εποχή κρίσεως διότι η ΕΚΤ έχει ε, λειτουργήσει θαραλέα, αλλά ήταν αναπόφευκτο ότι έπρεπε να το πράξει και σε περίοδο κρίσεως πρέπει να το πράξει μαζί και από κοινού με τις φορολογικές αρχές και τις ε, εθνικές αρχές, διότι πλέον δεν μιλάμε μόνο για ρευστότητα, αν και τα περισσότερα προβλήματα που έχουν οι χώρες πλην της Ελλάδος είναι θέματα ρευστότητος, αλλά ε, το όριο μεταξύ της ε, ε, ρευστότητος και της αξιο είναι πολύ λεπτό και ευέλικτο. Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικός ο λόγος αυτός ο οποίος υπάρχει και θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία της ΕΚΤ με ε, τις φορολογικές αρχές και ελπίζω ότι θα κατευθύνουν το πλοίο μας προς μια διαφορετική κατάσταση και όχι πλέον με την ομοφωνία η οποία απαιτείται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ και τώρα ερχόμαστε στον επόμενο μιλητή, τον Ρικάτο Καμπράλ. Έχετε λάβει τα βιογραφικά τους, οπότε δεν θα κάνω μια επίσημη ε, εισαγωγή. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που βρίσκομαι ενώπιον αυτής της Επιτροπής για να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Κρίση Δημοσίου Χρέους. Η μαρτυρία μου έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την προοπτική μου ως προς τη φύση της κρίσης σε σχέση με την αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα ήθελα να πω ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται σε μια κατάσταση αστάθειας και άρα η πλαισίωση και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ε, είναι ασυνεπές και επικίνδυνο. Η κρίση της Ευρώπης ως προς το ε, χρέος είναι μία κρίση ισοζυγίου πληρωμών και εξωτερικού χρέους. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι τα εξωτερικά ελλείμματα έχουν φτάσει σε επίπεδο χωρίς προηγούμενο σε σχέση με τα ισοζύγια πληρωμών τα στοιχεία 1, 2 και 3 δείχνουν ότι 12 χώρες ίσως έχουν επιπρόσθετο εξωτερικό χρέος. Ορισμένοι και πολλοί εμπειρογνώμενες θα μπορούσαν να θεωρούσαν ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα εξωτερικό χρέος της τάξης του 40% του ΟΕΠ. Πολλές χώρες βρίσκονται στο διπλό επίπεδο του 40% του ΟΕΠ ως προς το εξωτερικό χρέος. Πρόκειται για μία μη βιώσιμη πορεία εξωτερικού χρέους και τα προηγούμενα δείχνουν ότι το ε, χρέος, το εξωτερικό χρέος αυτών των χωρών θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν ε, προβεί σε προγράμματα για έξι χώρες, για την Ουγγαρία, τη Λετωνία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και βλέπουμε ότι πρόκειται για χώρες που είχαν πολύ υψηλά ελλείμματα ισοζυγίου εσόδων. Αυτό το βλέπουμε για την Ουγγαρία, την Λετωνία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. σε σχέση με αυτά τα ελλείμματα ισοζυγίου εσόδων. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν προαπαιτήσεις που σχετίζονται με το με τα έσοδα, μάλλον με τα εμπορικά ελλείμματα και με τα ελλείμματα ισοζυγίου εισοδήματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολύ υψηλές προαπαιτήσεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μειώσει αυτά τα δημοσιονομικά ελλείμματα σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όμως αυτά τα μέτρα είναι αντιπαραγωγικά. Για να κατανοήσουμε για θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι αυτός ο τύπος που ορίζει το, τις δανειοληπτικές ανάγκες μιας χώρας οδηγεί στον τύπο των μακροοικονομικών του 1 συν 3 ίσον 2 συν 2 για να ορίσουμε αυτά τα εμπορικά ελλείμματα καθώς και το έλλειμμα και τα ελλείμματα ισοζυγίου εσόδων ή εισοδήματος. Και σε αυτά τα πλαίσια τα μέτρα δημοσιονομικών, ε, τα δημοσιονομικά μέτρα δεν θα επιτύχουν όταν μιλάμε για μια καθοδική πορεία. Για παράδειγμα, το εμπορικό έλλειμμα της Πορτογαλίας το 2010 ήταν 6,5% του ΑΕΠ και 4,6% ε, του ΑΕΠ ήταν το ισοζύγιο, το έλλειμμα ισοζυγίου εισοδήματος. Γι' αυτό το πρόγραμμα προσαρμογής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα έπρεπε να σταθεί στο εμπορικό έλλειμμα καθαρά. Έτσι ώστε να δούμε τι αντιστοιχίες υπάρχουν. Επίσης το πρόγραμμα προσαρμογών θα έπρεπε να λάβει υπόψη ένα, μια ρεαλιστική αναδιάρθρωση χρέους. Βλέπουμε όμως ότι πρόκειται για χτυπήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Είναι σαν να χρησιμοποιούμε μία βαριοπούλα για να χτυπήσουμε ένα καρύδι. Μιλάμε δηλαδή για δραστικές μειώσεις οικονομικής δραστηριότητας και γι' αυτό δεν μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε το εμπορικό έλλειμμα το οποίο να βρίσκεται κοντά στο 6,5% του ΑΕΠ. Μιλάμε λοιπόν για μειώσεις σε σχέση με τις απαιτήσει δανειοδοσίας αυτών των χωρών. Επίσης, επειδή δεν λαμβάνονται υπόψη ε, σωστά τα ελλείμματα αυτά, βλέπουμε ότι ακολουθούμε μία ανωδική πορεία ελληματικών ισοζυγίων και όχι καθοδική. Έμπρακτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα μπορέσουν να επιλύσουν το πρόβλημα σε σχέση με, την, ε, με τις δραστικές μειώσεις που επιβάλλουν. Και οι ανάγκες δανειοδοσίας θα αυξηθούν. Επειδή λοιπόν ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες δανειοληψίας, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο δημόσιος τομέας. Επίσης, τα προγράμματα προσαρμογής δεν λαμβάνουν υπόψη την αναδιάρθρωση δημοσίου χρέους και δεν λαμβάνουν υπόψη το ισοζύγιο εσόδων. Γι' αυτό και η μόνη δικλίδα ασφαλείας για την μείωση του δημοσίου ελλείμματος θα ήταν να υπάρξουν πολλές βελτιώσεις στο εμπορικό ισοζύγιο και δεν θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πολιτική επαιτίας προς τις γείτονες χώρες. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε να κάνουμε με μια συνολική πολιτική ύφεσης. Το λιγότερο σημαίνει περισσότερο. Χρειάζονται λοιπόν στοχοθετημένες δραστηριότητες για να φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Η διαδικασία προσαρμογής είναι να ορίσουμε το εξωτερικό χρέος και να το σταθεροποιήσουμε το εξωτερικό χρέος των χωρών που έχουν υψηλές ανάγκες δανειοδότησης, έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε την οικονομική δραστηριότητα αυτών των χωρών. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, η εξωτερική προσαρμογή που χρειάζεται είναι της τάξης του 8% του ΕΕΠ. Και στην περίπτωση των ελλημάτων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες ε, δανειοδότησης σε σχέση με το εμπορικό έλλειμμα και το έλλειμμα ε, εισοδήματος, εξωτερικό έλλειμμα εισοδήματος. Έτσι θα φτάσουμε σε μια αποτελεσματική πολιτική. Επίσης, η πορτογαλική κυβέρνηση θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα, το δημοσιονομικό της έλλειμμα κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση με μια συγκεκριμένη φορολογική πολιτική η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια αναδιάρθρωση. Πιστεύω ότι μια πολιτική λοιπόν ε, φορολογικής υποτίμησης, fiscal devaluation, θα βοηθούσε έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η δημοσιονομική πολιτική. Για να έχουμε και μείωση του ΦΠΑ. Δεν πρέπει να προωθήσουμε την αύξηση αλλά τη μείωση του ΦΠΑ. Έτσι θα φτάναμε σε ένα 40% του ΑΕΠ στις χώρες της Ευρωζώνης από πλευράς ζήτησης θα πρέπει να επανισορροπήσουμε τους φόρους έτσι ώστε να έχουμε μείωση των τιμών στα εγχώρια προϊόντα και αυτό αφορά και τον τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών και του τομέα των υπηρεσιών, του τριτογενούς τομέα. Η αναδιάρθρωση του χρέους θα είχε σαν στόχο την μείωση των ε, ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έτσι ώστε οι περιφερειακές χώρες να είναι σε θέση από μόνες τους να βρεθούν εκ νέου, να μπουν εκ νέου στις αγορές. Και επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε ένα, ε, μία εξυγίανση των τραπεζών τύπου ΙΠΑ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Η τρέχουσα πολιτική είναι λανθασμένη και επικίνδυνη. Το πρόγραμμα προσαρμογής του Δούνου του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα βοηθήσει στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Πρόκειται για μια κατάσταση που οδηγεί στην αποδόμηση και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα οι περιφερειακές χώρες μπορούν να μειώσουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα εάν μπορούν να ε, βελτιώσουν τα εμπορικά τους ισοζύγια. Γι' αυτό η πολιτική ανταπόκριση στην κρίση σημαίνει ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε αυτές, αυτά τα ισοζύγια δεν θα πρέπει να ζητήσουμε ε, ρηξικέλευθες αλλαγές στο, σε, ολόκληρο, σε ολόκληρη τη διάρθρωση του οικονομικού και του, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να αντιμετωπίσουμε επί της ουσίας την, ε, κρίση χρέους, την δημόσια κρίση χρέους. Η οποία... Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα σε ένα γύρο ερωταπαντήσεων. Δεν ξέρω ποιος θέλει να θέσει ερωτήσεις. Συνήθως ε, προς το τέλος ε, έχουμε τους, ε, το γύρο ερωτήσεων, αλλά τώρα έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές, τους οποίους καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Σαπίρ μου είπε πάρα πολλά σχετικά με την διαφορά του προφίλ των χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσεως. Και αν κατάλαβα καλά τον κύριο Καπράλ, ε, θα ήθελε να υπάρξει μια διαφορετική κατεύθυνση ε, και αντιμετώπιση των ε, πληγέντων χωρών αλλά ουσιαστικά αυτό αναφέρεται στο πρώτο θέμα της συζητήσεως σήμερα. Ε, και βλέπουμε ότι ε, τα κράτη απομακρύνονται ε, με τον δε δραματικά βλέπουμε ότι και τα spreads θα αυξηθούν έχουμε ανησυχίες και στη συνέχεια με τη Γαλλία και προηγουμένως με την Ισπανία και την Ιταλία που θα χρειαστούν μεγαλύτερο τεραποσά επέμβαση στο 2012 οπότε εφόσον μιλάμε για μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να αποφύγουμε ε, μια διάλυση της Ευρωζώνης τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ο κύριος Σαπίρ ζήτησε επικοδομητική αντιμετώπιση ε, αντιλαμβάνομαι ότι η Τράπεζα της Αγγλίας προσπαθεί επιπλέον να προστατεύσει το δικό της νόμισμα και το EFSF όπως έχει καταρτιστεί δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες οπότε τι χρειάζεται, τι πρέπει να ενοποιήσουμε για να μπορέσει ο καθένας να διαδραματίσει το ρόλο που χρειάζεται. Τι θα γίνει με αυτά τα θεσμικά ε, όργανα. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να μας κάνετε μερικά πιο ακριβή σχόλια επί των θεμάτων. Όποιος από τους δυο σας, ο Αντρέ. Ναι, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια σε σχέση με το ρόλο του μηχανισμού ESFS. Πάντοτε βλέπω αντίφαση όταν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων λένε θα κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί για να επιλύσουμε την κρίση και πριν κάνουν πάρουν ανάσα μας λένε ότι το EFSF είναι 440 δις. Εμένα αυτά τα δύο δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι ισοδύναμα. Και όποιο βλέπει τι γίνεται στην Ευρωζώνη και ιδίω ε, ε, οι αγορές που παρακολουθούν τα πράγματα βλέπουν την αντίφαση μεταξύ των δύο αυτών φράσεων. Η μία έρχεται σε σχέση με την άλλη. Τι θα πει αυτό, οτιδήποτε χρειάζεται. Τελεία, δεν βάζεις αριθμό μετά από αυτό. Είσαι έτοιμος να κάνεις ό,τι χρειαστεί. Εάν όμως μετά βάζεις ένα περιορισμό, όπως είπα και πριν, αν περιορίζεις δίνοντας έναν αριθμό, πρώτον 440 δις και δεύτερον λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει ομοφωνία προτού αναλυφθεί δράση, αυτό πλέον αναιρεί το πρώτο κομμάτι. Και ναι, μεν χαιρετίζω αυτό το μηχανισμό και ο τελευταίο είμαι που θα πει ότι πρέπει να καταργηθεί. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό βήμα αυτό που έγινε, αλλά όσο εξελίχθηκε η κρίση φάνηκε ότι ήταν και ανεπαρκή ο μηχανισμό αυτό. Εξού και είπα και πριν ότι κατά την άποψή μου όταν κανεί έχει να αντιμετωπίσει μια κρίση και τέτοια φύση και τέτοιων διαστάσεων θα πρέπει σε αυτές τις λέξεις οτιδήποτε χρειαστεί να βάλεις περισσότερη αξιοπιστία. Άρα χρειάζεσαι κάτι διαφορετικό από το να αναφέρεις ένα ποσό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο ρόλος μιας κεντρικής τράπεζας, εκτός βέβαια αν πιστεύει κανεί ότι τελικά υπάρχει και ζήτημα φερικιότητας. Οπότε, και εκεί είπα ότι έκανα, κάνω τη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών. Thank you. Σας ευχαριστώ. Είπατε τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο βήμα είναι να ανασταλεί η εφαρμογή των προγραμμάτων που είναι σε ισχύ τώρα, διότι αυτό κάνει τις οικονομίες να πηγαίνουν προς τα πίσω και όχι προς τα εμπρός. Δεύτερον, συνιστώ να γίνουν ε, σημαντικές αλλαγές και δει στη φορολογική δομή, στη δομή της φορολογίας. Νομίζω ότι αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, ε, δεν μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την φορολογική δημοσιονομική υποτίμηση, fiscal devaluation. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο του EFSF, κατ' εμέ ξέρω γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο μηχανισμός, δημιουργήθηκε για να ανταποκρίνεται σε κάποια κατεπήγοντα περιστατικά, σε καταστάσεις ανάγκης, αλλά η στόχη και η δομή του EFSF δεν είναι επαρκώς ε, ξεκάθαρη αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο κατ' εμέ χρειάζεται στην Ευρώπη είναι ε, να έχουμε ένα καθεστώς πραγματικής resolution των προβλημάτων χρέους. Uh, Εγώ έχω να κάνω ένα ερώτημα προς τον κύριο Σαπίρ που είπε ότι ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας εν καιρό κρίσης θα πρέπει να είναι διαφορετική. Δηλαδή δεν μιλάμε για, δεν μιλάμε για κανονικές συνθήκες. Είπατε και για τη ΦΕΝΤΕ, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Γιατί μιλάτε τελικά για τη λεγόμενη ποσοτική ελάφρυνση, αυτό το quantitative easing που εφαρμόζουν στις ΗΠΑ ή μιλάτε συγκεκριμένα για την ΕΚΤ. Επειδή η Ευρωζώνη δεν πληρεί τα κριτήρια της ε, περιοχής του κοινού νομίσματος, άρα είναι κάτι διαφορετικό από τη ήπα και είναι κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει η έκτα να ξεπεράσει αυτά που κάνει η ΦΕΔ, επαναλαμβάνω, εν καιρό κρίσης. Να σας απαντήσω ε, λέγοντας ότι ουσιαστικά ε, δεν μίλησα ε, πολύ συγκεκριμένα. Γενικώς το ανέφερα. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω πλήρως και θα το συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της ακρόασης. Καταλαβαίνω πλήρως, επαναλαμβάνω, τους περιορισμούς, θα έλεγα τους πολιτικούς περιορισμούς. Κατανοώ απόλυτα το πώς η ΕΚΤ δημιουργήθηκε και το πώς δημιουργήθηκε και η Ευρωζώνη. Καταλαβαίνω και τι είδους ε, πολιτικό συμβόλαιο έχει συναυθεί τελικά και ποια είναι η ευθύνη του καθενός πρωταγωνιστή στην Ευρωζώνη, κυβερνήσεις και κεντρικές ε, τράπεζες. Ο καθένας έχει το ρόλο του να διαδραματίσει. Αυτό το συμβόλαιο έχει παραβιαστεί κατά κάποιο τρόπο λόγω της συμπεριφοράς ορισμένων χωρών. Αλλά για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας θέλω να σας πω ότι έχοντας ε, εργαστεί διαμαρκών στην Ευρωζώνη και πριν ε, εισαχθεί το ευρώ, δεν είμαι αρχιτέκτονας, αλλά τέλος πάντων συμμετείχα στις συζητήσεις επί του σχεδιασμού της Ευρωζώνης. Νομίζω λοιπόν ότι μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαμε σκεφτεί. Και ένα από τα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι δεν αντιληφθήκαμε στην πλήρη τους διάσταση ήταν η ιδέα ότι χώρες, και αυτό είναι η ιδιαιτερότητα της Ευρωζώνης, χώρες που είναι στην Ευρωζώνη μπορούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ό,τι αφορά το χρέος. Δεν το φανταστήκαμε, δεν, δεν, δεν το σκεφτήκαμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. δεν σκεφτήκαμε ότι κάποιο ναι μεν ε, μπαίνει σε μια ζώνη κοινού νομίσματο και σίγουρα αυτό του δίνει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά δημιουργεί και κάποιε προποθέσει και κάποιου όρου. Οι αγορέ ενδεχομένω κάποια στιγμή χάσουν την εμπιστοσύνη του στα κρατικά ομόλογα ορισμένων χωρών. Αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Κάναμε διάφορα πράγματα. Είχαμε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο, είχαμε το σύμφωνο σταθερότητα αλλά αυτό και τα πιθανά προβλήματα αφαιρεγκιότητας πάυσης πληρωμών, στάσης πληρωμών μάλλον, δεν τα αντιμετωπίσαμε. Δεν σκεφτήκαμε τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση κρίσης, με άλλα λόγια. Σχεδιάσαμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να ανταποκρίνεται υπό κανονικές συνθήκες, αλλά η δύσκολη θέση αυτών των δυόμιση τελευταίων ετών έγκυται ακριβώ ότι πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε μια κατάσταση κρίσης. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο συνάδελφο ε, Καθηγητή Καμπράλ για την οικονομική πλευρά, τη χρηματοπιστωτική πλευρά. Στη συνθήκη του Μαστρίχτ τίποτα δεν υπάρχει το οποίο να έχει να κάνει απευθεία με τα οικονομικά θέματα. Γίνεται όσο τα φορολογική βιωσιμότητα, fiscal ε, sustainability. Και εκεί πάλι δεν κάναμε πολλά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ασχοληθήκαμε με το λεγόμενο financial sustainability, την οικονομική βιωσιμότητα, το ιδιωτικό χρέος. Και αυτό βέβαια γιατί η συνθήκη του Μαστρίχτη ήταν πριν από 20 χρόνια. Και όπως συμβαίνει συχνά, κοίταζε προς τα πίσω, δεν κοίταζε προς τα εμπρός. Έναν κόσμο δηλαδή που θα υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, όπου θα υπάρχει μεγάλη οικονομική χρηματοπιστωτική διασύνδεση, που υπάρχουν χώρες που συσσωρεύουν κρατικό χρέος, όλο αυτό το φαύλο κύκλο στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Έχουμε τις, τα, τα ομόλογα που είναι αδύναμα, οι τράπεζες είναι αδύναμες, όλος αυτό ο φαύλος κύκλος. Αυτό δεν ε, το λάβαμε υπόψη στην συζήτηση που κάναμε. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε λοιπόν το πλαίσιο που έχουμε, το επικαιροποιήσουμε, αλλά στο μεσοδιάστημα, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, θα πρέπει αυτό το πλαίσιο που έχουμε να το εφαρμόσουμε με ευελιξία. Σίγουρα έχει τίμημα αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι χειρότερη οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική. Σας ευχαριστώ. Okay, if you could please put the θα ήθελα να βάλετε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Έχω ένα ε, σχόλιο και δύο παρατηρήσεις. Οι ε, αρχηγοί κυβερνήσεως θεωρούν ότι ε, δεν κινούνται αρκετά γρήγορα να καθησυχάσουν τις αγορές. Βλέπουμε όμως ότι οι εμπειρογνώμονες δεν συμφωνούν επί του πρακτέου. Και όταν το τον έναν επιστήμονα ο οποίος έχει πάρει βρεβείο Νόμπελ Οικονομικών που είπε πώς μπορεί να λύσουμε την ε, κρίση βλέπω ότι δεν είναι εύκολο να καταλήξει κανείς σε μία σαφή εικόνα και η, ε, ε, πρώτη μου ερώτηση είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να υπάρχει μία αξιόπιστη βάση. Δεύτερον, Οντρέ, συμφωνώ ότι θα έπρεπε να θεωρούμε ότι η ΕΚΤ είναι ο δανειοδότης τελευταίας διαφυγής χωρίς περιορισμούς. Αλλά αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο κίνδυνο δημοκρατικής νομιμοποίησεως, διότι αν δεν υπάρχει ο αν δεν υπάρχει ομοφωνία τότε οι φορολογούμενοι είναι όμοιροι ορισμένων αποφάσεων και ε, ποιος μου λέει ότι οι χώρες οι οποίες είναι ακόμη σε καλή οικονομική κατάσταση αλλά ε, θα εγγυηθούν ενδεχομένως αυτά τα δάνεια θα χάσουν την ε, θέση τους σαν χώρες με τριπλό αλφα και θα καταλήξουμε στην Ευρωζώνη χωρίς να υπάρχει καμία χώρα με τριπλό αλφα αξιολόγηση και προς τον καθηγητή Καμπράλ. Από ό,τι κατάλαβα για την κριτική την οποία εξασκήσατε για την πολιτική βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι προφανές ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε σε σχέση με την περισσυνή αντί να βελτιωθεί. Και είναι κάτι το οποίο δεν είχε σκεφτεί ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευθύνη ουσιαστικά είναι στο, Ευρω... στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εάν λοιπόν συστήματα έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν, γιατί τώρα δεν λειτουργούν. Και πόσο δυσχερής θα γίνει η κατάσταση ε, το διαπιστώνω διαβάζοντας ε, μία έκθεση της Commerzbank όπου λέει ε, ότι η Γερμανία του χρόνου θα έχει 0,8 η Γαλλία 0 και η Ισπανία 0,3% δηλαδή βλέπετε ότι οι μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης δεν, δεν θα έχουν ή καθόλου ανάπτυξη ή μία ελάχιστη ανάπτυξη. Οπότε το ερώτημα είναι, εάν ακολουθήσουμε την πρότασή σας κύριε Καμπράλ, ε, εάν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τα ελλείμματα. Thank you. Um, Κλείστε και το μικρόφωνο σας. Thank you ως προς τα μέτρα λιτότητας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν αντιτάσσομαι στη λιτότητα καθεαυτή. Απλώς θεωρώ ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι λογικά. Οι πολιτικές αυτές. Έχουμε μία εξίσωση και το πακέτο αυτό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προσπαθεί να αλλάξει τους όρους αυτής της εξίσωσης, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει η εξίσωση από την αριστερή πλευρά χωρίς να αλλάξει η δεξιά πλευρά. Δηλαδή, ως προς το εμπορικό ισοζύγιο και το έλλειμμα που υπάρχει στο ισοζύγιο εσόδων. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι αν προσπαθήσετε να πιέσετε την αριστερά πλευρά, πιέζετε τα πάντα. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Θα μειώσουμε το έλλειμμα εάν μειώσουμε το εμπορικό ισοζύγιο. Αυτό σας είπα. Και το τρέχον πακέτο είναι ζημιογόνο για πλεονασματικές χώρες όπως η Γερμανία, για χώρες με πλεόνασμα, διότι όλα μπαίνουν στο εμπορικό ισοζύγιο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτές τις 12 χώρες. Θα πρέπει να αλλάξουμε από ε, ισοζύγιο, ελληματικό ισοζύγιο σε πλονασματικό ισοζύγιο ως προς το εμπορικό του ισοζύγιο και μόνο έτσι θα μπορέσει να επιτευχθεί κάτι. Δεν ξέρω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ορίζουν μια τέτοια πολιτική αυστηρής λιτότητας. Δεν είναι ποτέ εύκολο να ανταποκριθεί κανείς σε μια κατάσταση κρίσης. Δυστυχώς οι επικεφαλείς έχουν συγκρουόμενες απόψεις. Χρησιμοποιούν σύμβουλους, το ένστικτό τους και πολλές φορές ε, σφάλουν. Ας ελπίσουμε ότι έχουν φτάσει στις καλύτερες δυνατές λύσεις. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε Τρία είναι τα καλά πράγματα, ε, προσθέτει γερμανικά. Δηλαδή, πρέπει να ε, αναλύσετε τις εναλλακτικές λύσεις και να ξεχωρίσετε τις καλές από τις κακές. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με την βέλτιστη δυνατή οικονομική διακυβέρνηση, αλλιώς δεν γίνεται. Θα ήθελα και εγώ να σας απαντήσω σε σχέση με τη δημοκρατική νομιμότητα και την αρχή της ομοφωνίας. Νομίζω ότι θα επανέλθει στο δεύτερο τμήμα των συζητήσεών μας, διότι μας οδηγεί στο μέλλον, στην, ε, στην φορολογική ολοκλήρωση, στη φορολογική ένωση και πώς θα επιτευχθεί. Πολλές φορές ακούω επικρίσεις για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα η Γερμανία κατά την κρίση. Και θα πρέπει να πω ότι δεν συμμερίζομαι αυτές τις επικρίσεις. Καθόλου δεν τις συμμερίζομαι. Θεωρώ ότι η Γερμανία συνέβαλε σημαντικά και δραστικά αν θέλουμε να κάνουμε μία σύνδεση με αυτό που είπαμε ε, πριν. Και δούμε και την ε, εξέλιξη, την ιστορική εξέλιξη πριν από το ευρώ. Η Γερμανία είχε προσυζητήσει αυτά τα θέματα για το συσχετισμό μεταξύ νομισματικής ένωσης και φορολογικής ένωσης. Εκεί είχαν πρωταρχικά γίνει οι συζητήσεις. Και δυστυχώς η νομισματική ένωση δημιουργήθηκε με μία μόνο χώρα, με μία μόνο χώρα, από τη Γερμανία. Μόνο η Γερμανία ε, αποποιήθηκε την κυριαρχία της. Καμία άλλη χώρα. Καμία άλλη χώρα δεν διέθετε αυτή την κυριαρχία. Μόνο η Γερμανία την διέθετε και την απαρνήθηκε. Το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε μία διαφορετική επιλογή. Δηλαδή ήθελε να κρατήσει την νομισματική της κυριαρχία. Αλλά το Μάρκο είχε πραγματική κυριαρχία. Και οι άλλες χώρες κέρδισαν μέρος της κυριαρχίας που διέθετε μόνο η Γερμανία. Και ε, το δράμα έγκυται στο ότι μόνο στη Γερμανία είχαν προσυζητηθεί αυτά τα ζητήματα που πέρασε δηλαδή από το γερμανικό μάρκο στο ε, ευρώ. Δηλαδή υπαναχώρησε σε σχέση με το γερμανικό μάρκο όπου είχε πραγματική κυριαρχία. Οι άλλες χώρες δεν είχαν να καταβάλουν αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή οι άλλες χώρες είχαν ένα δωρεάν αντάλλαγμα, αν θέλετε. Και αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Δεν είχαν να αποποιηθούν οι άλλες χώρες κάτι. Η νομισματική ένωση θα πρέπει να είναι μια σύμβαση στο μέλλον, όπου κάθε χώρα υπαναχωρεί ως προς κάτι για να συμμετέχει στη σύμβαση αυτή. Τώρα, μελλοντικά, πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε μία νέα συνθήκη η οποία θα διορθώσει τα σφάλματα του παρελθόντος που θα βελτιώσει δηλαδή την ε, τελευταία συνθήκη. για να μιλήσουμε για ποιο μέρος της εθνικής κυριαρχίας θέλουν να αποποιηθούν και άλλες χώρες. Διότι σε άλλες χώρες δεν έχει καν αρχίσει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή η μελλοντική νομισματική ένωση θα πρέπει να είναι αυτό που ήταν για τη Γερμανία τα τελευταία 12 χρόνια η οποία αποποιήθηκε την εθνική της κυριαρχία για το κοινό καλό. Όσο νωρίτερα αρχίσει η συζήτηση, τότε θα φτάσουμε σε μία πιο εξισορροπημένη νομισματική ένωση με όλα τα στοιχεία που λείπουν αυτή τη στιγμή. Και δεν θα υπάρχει θέμα δημοκρατικής νομιμότητας, διότι θα υπάρχουν όλα τα θεσμικά στοιχεία ενσωματωμένα. Τώρα δεν υπάρχει πλήρης νομιμότητα γιατί δεν έχουμε μια συνθήκη η οποία να υποστηρίζει αυτές τις δράσεις. Και όμως πρέπει να δράσουμε για να επιλύσουμε την κρίση. Και το τελευταίο ερώτημα. Um, Και ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τις τελευταίες εβδομάδες έχω συζητήσει με διάφορους επενδυτές ε, παγκόσμιους επενδυτές που θέλουν να συμμετάσχουν ε, στην Ευρωζώνη και νομίζουν ότι αν καταλάβουν τι γίνεται θα μπορούσαν να διαθέσουν κάποια κονδύλια. Και ένα από αυτά που μου έχουν επισημάνει είναι ότι υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας ενός ε, ειδικού οχήματος του EFSF και δεν ξέρουν κατά πόσο είναι το σωστό όχημα αυτό, γιατί ουσιαστικά από τις αγορές ε, εισπράττει κάποια χρήματα και όχι από τα κράτη-μέλη. Περιμένουν λοιπόν ε, από τις αγορές. Όταν λοιπόν ασκηθεί μόχλευση, και αυτό ακούμε αυτή τη στιγμή στον τύπο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βλέπουμε να ανησυχούν οι επενδυτέ Όταν η Τράπεζα τη Αγγλίας κάνει κάποιε δηλώσει για αυτή την ε, ποσοτική ελάφρυνση, ε, δηλαδή ουσιαστικά ε, το να τυπώσουν χρήμα, οι επενδυτέ δεν καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν πως αυτό το όχημα τελικά μπορεί να είναι αποτελεσματικό και να κάνει και το ίδιο πράγμα. Ποιο είναι το ερώτημά μου. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να πείσουμε τις αγορές, άρα και τους παγκόσμιους επενδυτές, ότι αυτό το όχημα εντός αγωγικών μπορεί και λειτουργεί. Θέλει να απαντήσει πρώτος. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι το EFSF, ή τέλος πάντων η δομή που έχει παντων η οποία έχει φτιαχτεί, δεν είναι ξεκάθαρη, υπό μία έννοια. Ήταν ε, κάτι το οποίο δημιουργήθηκε σε κατάσταση, σε μια περίπτωση ανάγκης βλέπουμε ότι έχει το back office στην Ευρωπαϊκή Τρική Τράπεζα. Έχουμε ε, το Γραφείο Διαχείρισης του Χρέους, το οποίο δρεύει στη Γερμανία. Λέει ότι έχει ε, υπαλλήλους, αλλά στο καταστατικό αναφέρονται μόνο 19 υπάλληλοι και είναι ε, υπεύθυνο για 440 Solid construction. δις. Νομίζω λοιπόν ότι η μόχλευση προσθέτει σύγχυση και περιπλοκές και ίσως θα πρέπει να σας απασχολήσει ποιες εναλλακτικές, ποιες καλύτερες εναλλακτικές υπάρχουν. Ο Αντρέ, ευχαριστώ. Εγώ νόμιζα ότι θα πρέπει να δούμε το EFSF ε, στο τι κάνει συγκεκριμένα. Ο αρχικός του στόχος πράγματι ήταν να εργάζεται χέρι με χέρι με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε κοινά προγράμματα ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Δουνουτού στην Ευρωζώνη. Όπως συζητήσαμε, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία. Αυτά είναι τα τρία ε, προγράμματα. Και είναι το σκέλος που χρηματοδοτεί το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, αν θέλετε. Δηλαδή συνεργασία με το Διαθέσιμο Νομισματικό Ταμείο σε χώρες για τις οποίες έχουν καταρτιστεί αυτά τα προγράμματα εντός της Ευρωζώνης. Για μια τέτοιου είδους δραστηριότητα πιστεύω ότι το EFSF δεν έχει πρόβλημα. Μπορεί να τα καταφέρει, εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα, καμία δυσκολία. Τώρα ε, λέμε ότι ίσως πρέπει να είναι μόνιμος ο μηχανισμός, άρα που η FSF θα λέγεται ESM λοιπά. Δεν υπάρχει όμως ακόμη ομόφωνη, αλλά σε ό,τι αφορά την κατασκευή του και αν ένας επενδυτής ε, θέλει να βάλει τα χρήματά του στο EFSF, εγώ δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Αν εγώ ήμουν επενδυτής, υπό την έννοια αυτή δεν θα έβρισκα ότι το EFSF ε, δεν τα καταφέρνει καλά, δεν έχει σχεδιαστεί επαρκώς για να φέρει σε πέρα στο ρόλο αυτό. Το μόνο πρόβλημα ίσω είναι η ομοφωνία, ότι είναι ανάγκη να υπάρχει ομοφωνία για κάποιο πρόγραμμα, κάτι που δεν ισχύει ξεκάθαρα για το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το EFSF, εδώ μιλάμε για ένα νέο ρόλο. Για, μιλάμε για ένα βελτιωμένο, ένα νέο EFSF. Ένα μηχανισμό που το EFSF τώρα αναλαμβάνεται, εκπαιρεώσει κάποια καθήκοντα τα οποία κανονικά θα έπρεπε να επιτελεί μια κεντρική τράπεζα. Και σε αυτό το σημείο πράγματι και εγώ έχω κάποιες δυσκολίες να αποδεχθώ κάτι τέτοιο. Γιατί αν είχαμε σχεδιάσει το σύστημα καλύτερα, μπορώ να σας πω ότι τότε αυτή την ευθύνη, αυτή την αρμοδιότητα εγώ θα την είχα δώσει στην κεντρική τράπεζα. Είναι σαν να έχουμε ένα σταυροδρόμι ή τέλος πάντων μια διάβαση ανισόπεδη, ένα roundabout και εκεί γίνονται κάπως μπερδεμένα τα πράγματα. Το θέμα είναι να δούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ EFSF και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άπαξ και υπάρχει το βελτιωμένο EFSF, το έκτα e κατά μία άποψη βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Κατά την άποψή μου η άποψη αυτή είναι ακραία και δεν είναι βιώσιμη κάτε με, για τους λόγους που προανέφερα. Το ύφεσαι δεν μπορεί, κατά την άποψή μου πάντα, να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου την Κεντρική Τράπεζα. Μπορεί να έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο, ακριβώς λόγω αυτής της δυσκολίας αυτό το ε, σύνορο μεταξύ ρευστότητας, φερεγγιότητας. Αυτό που είναι σήμερα ένα πρόβλημα ρευστότητας φοβούμαστε ότι μπορεί να γίνει πρόβλημα φερεγγιότητας στο μέλλον. Οπότε μπορεί να ανησυχεί τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τη στηρίζουν κυβερνήσεις και τα Υπουργεία Οικονομικών και πώς και πόσο. Αυτό είναι ένα θέμα για του κεντρικού τραπεζίτε σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι όλο που εγώ θα ήθελα για το EFSF. Όχι να υποκαταστήσει πλήρως την Κεντρική Τράπεζα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Νομίζω ότι μας δώσατε πολύ τροφή για συζήτηση. Θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ και θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον Γιούργεν Στάρκ. Μετά θα περάσουμε στον Ζερόμ Κρέλ. Παρακαλώ, Γιούργεν Στάρκ, είστε ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής αυτής. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και μπορώ να συζητήσω μαζί σας θέματα ε, οικονομικής διακυβέρνησης. Είχα τον πειρασμό να επέμβω και στον πρώτο γύρο της συζήτησης γιατί ήδη πολλά ελέγχθησαν για τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας αλλά μπορούμε ίσως να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και στη συνέχεια. Θα ήθελα όμως τώρα στα λίγα λεπτά που έχω διαθέσιμα να αναφερθώ στα τρία θέματα τα οποία είναι προσυζήτηση σήμερα. Την εφαρμογή της, του πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης, το μακροπρόθεσμο, τις μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις στην οικονομική διακυβέρνηση και τα ευρωμόλογα. Καταρχήν ε, θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ σαν Επιτροπή ε, που υπερψηφίσατε το six pack τις έξι οδηγίες και κανονισμούς διότι μπορέσετε κατά αυτόν τον τρόπο να ενισχύσετε την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει η βούληση ε, να αντιμετωπίσετε ορισμένες αδυναμίες οι οποίες απεκαλύφθησαν σαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Χρειάζεται λοιπόν ένα πιο ισχυρό πλαίσιο από αυτό που είχε προτείνει αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πρόοδος οφείλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο ε, εξασκεί την εξουσία του για μια πιο ευρωπαϊκή και υπερεθνική προσέγγιση το, της οικονομικής διακυβέρνησης. Το θέμα είναι εάν πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες στα θέματα της φορολογίας για να μπορέσει να προωθηθεί η, ε, η ανάκαμψη στην Ευρώπη και τώρα βλέπουμε ότι όσον αφορά την ε, πολιτική σταθερότητος υπάρχει ε, μια νέα αναμόρφωση η οποία εφαρμόζεται στις ε, χώρες της Ευρωζώνης. Επίσης σημαντικό και ενισχυμένο από το Κοινοβούλιο είναι το θέμα της στατιστικής διακυβέρνησης που είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την ε, παρέμβαση στην αγορά. Όσον αφορά το πλαίσιο της μακροοικονομικής ε, εποπτείας, το πλαίσιο αυτό είναι πολύ σημαντικό και έπρεπε να προσθεθεί εις ε, τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι ο πίνακας βαθμολόγησης, το scoreboard, είναι επίσης πολύ σημαντικό διότι επιτρέπει επιτρέπει να εντοπίσουμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες θα παρεμποδίσουν τη χρηστή λειτουργία της νομισματικής ένωσης και ε, το scoreboard αυτό ε, φυστά την ε, προσοχή στις μακροοικονομικές ανισορροπίες ήδη από την αρχή. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Αλλά Δυστυχώς και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο αλλά ε, υπάρχει ακόμη μεγάλη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την εφαρμογή ε, και ε, την η αποτελεσματικότητα των μεσών εξαρτάται από την εφαρμογή τους όχι μόνο κατά γράμμα αλλά και ως προς το πνεύμα και γι' αυτό μπορέσαμε να αποκομίσουμε τις ε, εμπειρίες ε, που είχαμε μέχρι τώρα. Θεωρούμε ότι καταρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταρτίζει σωστές συστάσεις και στο Συμβούλιο να εξασκείται μία πίεση μεταξύ των ομολόγων και διάφοροι τομείς που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας αυτής ενισχύουν ότι την ανησυχία μας για το μεγάλο κίνδυνο της εφαρμογής και γι' αυτό η ε, ΕΚΤ λυπάται διότι ένα βασικό θέμα το οποίο πρότεινε δηλαδή μεγαλύτερη ε, αυτοματισμό και την ε, την ανάστροφη ε, ενισχυμένη πλειοψηφία δεν επετέύθη παρά μερικώς. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τα μέσα που διαθέτουμε, τον οικονομικό διάλογο για να εφαρμοστεί η ε, πειθαρχία στις αγορές ε, και να εξασκείται ε, πίεση προς τους ομολόγους και στη συνέχεια για να μπορέσει να υπάρξει η εποπτεία και να εξασκηθεί και η κοινοβουλευτική πίεση αλλά νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν και αυτό πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία εποπτείας και όλοι πρέπει να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτό σημαίνει να ε, διατυπωθεί εσωτερικά τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα διότι υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες δεν έχουν ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις της Ευρωζώνης και της Νομισματικής Ένωσης και ορισμένες παρεμβάσεις ξεκίνησαν με μεγάλη καθυστέρηση στην ε, ε, Νομισματική Ένωση. Βέβαια πρέπει να υπάρχουν και άλλες μετατοπίσεις ως προς τις αρμοδιότητες. Ο ζωμόνε που πολλές φορές έχει αναφερθεί ε, στο Κοινοβούλιο είχε τονίσει ότι υπάρχουν όρια στο συντονισμό διότι υπάρχουν όρια στη συζήτηση που δεν οδηγεί σε μία απόφαση και οι αποτελεσματικές αποφάσεις ε, ε, δεν μπορούν να γίνουν με ενδιαφέρους, να ληφθούν με ενδιαφέρουσες αλλά ατέρμονες συζητήσεις και αυτό με οδηγεί στην σύστασή μου ότι χρειάζεται να υπάρξει νέας ποιότητος διακυβέρνηση βάσει του πακέτου το οποίο έχει συμφωνηθεί και χρειάζεται μια πραγματική οικονομική ένωση και μία πρόοδος να εφαρμοστεί η πολιτική ένωση, δηλαδή η λύση είναι περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη Ευρώπη και φαντάζομαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει την ρήτρα αναθεώρησης για να προβεί σε αυτές τις βελτιώσεις διότι κατά τη γνώμη μου χρειάζεται ε, ε, εποπτεία μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και μία μετακίνηση της ε, κυριαρχίας προς το ευρωπαϊκό επίπεδο με μεγαλύτερες εξουσίες και μεγαλύτερους ε, περιορισμούς στην πολιτική ε, εθνικού προπολογισμού. Δηλαδή να μπορεί κανείς να καταρτίζει μακροφορολογικά κούσους στόχους και ε, να υπάρξει μία ουσιαστική και συνολική ανάταξη τη της συνθήκης για να επιλύσει κανείς και το θέμα της ε, δημοκρατικής νομιμοποίησης που φύγει προηγουμένως όχι μόνο στο, στην Ευρώπη αλλά και στα εθνικά κοινοβούλια. Και ο ακρογωνιαίος λίσθος αυτής της μεταρρύθμισης είναι ε, να υπάρξει μεταρρύθμιση που να επιτρέψει ε, το 3% του ΑΕΠ και να μπορέσουν μπορέσουν όλες οι κυβερνήσεις ε, της Ευρωζώνης να συμμορφωθούν και στους επόμενους προπολογισμούς ορισμένες αποκλήσεις από τους στόχους θα μπορούν αυτομάτως να διορθώνονται χωρίς καμία διακριτική ευχέρεια και θα χρειαστεί να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν οι ρόλια, ε, τα μέτρα αυτά και να συμπεριληφθούν και στα εθνικά συντάγματα. Ε, πρέπει λοιπόν τα μακροοικονομικά προγράμματα που λαμβάνουν υπόψη ε, την παρέμβαση ε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης ε, να επεμβαίνουν για να αποφευθεί η χρεοκοπία και θα υπάρχουν ανεξάρτητες δημοσιονομικές αρχές που υπάρχουν ήδη σε ορισμένες χώρες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής θα χρειαστούμε ένα αντίστοιχο οργανισμό με σαφή εντολή και τις δυνατότητες να εφαρμόσει τους φορολογικούς κανόνες κατά τρόπον ώστε να καταρτιστεί ένα ευρωπαϊκό γραφείο προϋπολογισμού που θα αποτελέσει τον πυρήνα αυτού που αργότερα θα οδηγήσει βαθμιαία σε ένα ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών. Είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ σοβαρά. Και έρχομαι τώρα στο τελευταίο μου θέμα, την έκδοση ευρωμολόγων. Κατά τη γνώμη μου, για να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση ε, που είναι κάτι απαραίτητο, μην νομίζετε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση που θα λύσει αυτή την κρίση και θα αποφύγει μελλοντικές ε, μέσω της εκδόσεως των ευρωμολόγων διότι η κατάσταση ε, των χρεών οφείλονται σε απαράδεκτες φορολογικές πολιτικές και χρειάζεται η εφαρμογή ε, των ε, προσεκτικών και βιωσίμων φορολογικών πολιτικών και κινήτρων που θα επιτρέψουν μακροπρόθεσμα την επίλυση του προβλήματος. Το γεγονός ότι η αγορές ζητούν υψηλότερες αποδόσεις για να χρηματοδοτήσουν τις χώρες είναι μία πίεση να, να ε, υποκινήσουν τις χώρες αυτές να διορθώσουν τα οικονομικά τους αλλά δεν έπρεπε να υπάρχουν καν αυτές οι αποδόσεις και θα πρέπει να υπάρχει μια ανακατανομή του κόστους της τωρινής κράσεως και δεν είναι προφανές ότι τα ευρωομόλογα θα βοηθήσουν στην επίλυση της κρίσεως. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν και εδώ μιλώ προσωπικά τα ευρωομόλογα δεν επιλύουν την, ε, την κρίση των κρατών την οποία να αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη παρουσίαση από τον Ζερόμ Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές. Ε, με τιμά ιδιαίτερα που μου δώσατε τη δυνατότητα να σας μιλήσω σήμερα και να σας ε, δώσω κάποιες από τις δικές μου σκέψεις σε σχέση με το νέο θεματολόγιο των πολιτικών μεταρρυθμίσεων, κάτι που σας απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς ε, θα σας πω το εξής. Νομίζω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο κινδύνους ε, μετάδοσης και με μία άλλη μετάδοση. Πρώτος κίνδυνος ε, είναι η δυσπιστία, η έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει σε κάποια ε, κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και τελικά η έλλειψη εμπιστοσύνης που θα μπορούσε να είναι γενικότερα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Δεν ξέρω πώς θα πούμε το νέο μηχανισμό, η FSM, η FSF, η ESM, ευρωομόλογα, γιατί θα μιλήσουμε δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε μια λύση ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη και προς το ευρώ και προς τα θεσμικά όργανα. Μια άλλη ε, μετάδοση ε, είναι των κακών συμπεριφορών. Πρέπει να πούμε ότι κάποιες κυβερνήσεις δεν συμπεριφέρθηκαν με τον σωστό τρόπο ε, στη διάρκεια της κρίσης. Και για χρόνια γνωρίζαμε, για παράδειγμα, ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε πρόβλημα με τα δημόσια οικονομικά. Άρα είναι λογικό να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο κινδύνους ε, μετάδοσης, αλλά μπορεί να έχουμε και μία φορολογική συρρήκνωση ταυτόχρονα. Και αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα, γιατί στην παρούσα κρίση αναδείχθηκαν κάποιοι νικητές και κάποιοι τιμένοι. Οι τιμένοι είναι, παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένοχη όμως. Υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, που ε, είναι ε, μεταξύ των τιμένων χωρίς να είναι και τόσο υπεύθυνοι. Υπάρχουν και άλλες χώρες, θα ε, δούμε τη Γαλλία, ε, αν δείτε τα επιτόκια, θα δείτε ότι είναι, ε, παραδείγματος χάρη, αυξημένα πολύ για την Ελλάδα τα επιτόκια, ενώ για τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία είναι πολύ πιο χαμηλά. Και αυτό αφήνει κάποια περιθώρια ελιγμών, ώστε να μπορέσουν οι χώρες αυτές να δείξουν αλληλεγγύη. Πρέπει λοιπόν την επόμενη εβδομάδα να βρεθεί λύση για να σταματήσει αυτή η κρίση. Επειδή όμως μου ζητήθηκε να μιλήσω για την οικονομική διακυβέρνηση, νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητα των δικών μα ε, θεσμών να αντιμετωπίσουν στο μέλλον χώρε που δεν συμπεριφέρονται σωστά. Δεν νομίζω όμω ότι μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο αξιότιμο συνάδελφο ε, μόλι πριν από λίγο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε νέου θεσμού. Μα έχετε δείξει ήδη ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση, διότι κατά την άποψή μου κάνατε καταπληκτική δουλειά με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που έχετε συμπεριλάβει στο μηχανισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πλέον παρακολουθούνται αυτές οι ε, διαφορές, οι τόσο μεγάλες διαφορές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό το οποίο με εντυπωσίασε είναι ότι μεταξύ των ε, τροποποιήσεων 27 Σεπτεμβρίου μας λένε πλέον ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες αποτελούν, συνιστούν αυτόματα έλλειμμα θα μπορούσαν να είναι όμως και πλεόνασμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για χώρες που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι οι μόνοι κακοί μαθητές. Αλλά για να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, νομίζω ότι πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτη, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δημοκρατία και όχι την απλούστευση για να μπορέσουμε να βαθμονομήσουμε, να μετρήσουμε τη μεταρρύθμιση πολιτικής. Έχουμε του ε, συναδέλφους ε, Κόπιτς και και οι οποίοι έχουν ε, αναφέρει κάποιους κανόνες, ότι πρέπει οι φορολογικοί κανόνες να είναι καλώς ορισμένοι, διαφανείς, απλοί, ευέλικτοι κτλ. Δεν νομίζω όμως ότι και αυτό. Είμαστε σε ένα πολύπλοκο κόσμο. Ίσως λοιπόν χρειάζονται και πολύπλοκοι, όχι απλοί κανόνες. Απλά θα πρέπει να τους έχουμε ορίσει καλά και θα πρέπει να τους ελέγχουν η ενδιάμεση ή ο ίδιος ο κόσμος. Και ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να παρακολουθεί, να ελέγχει ε, την υλοποίηση αυτών των κανόνων. Θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη δημοκρατική αρχή όταν κοιτάμε τους φορολογικούς κανόνες. Κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι συζητούμε εδώ τις αλλαγές, τα δημόσια οικονομικά στις διαφορετικές αυτές χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Πρέπει να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της φορολογικής πολιτικής και πραγματικά δυσκολεύομαι με το γεγονός ότι πολλές συζητήσει για τη παρολική πολιτική χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη επισιοδοξία. Και τελικά παίρνουν ε, το ρίσκο να μην εμπιστεύεται ο κόσμο στην κυβέρνησή του τελικά. Γιατί η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία τελικά δεν εφαρμόζει τι σωστέ πολιτικέ και φοβούμε ότι δεν θα υπάρχει πιστοσύνη ούτε και προ του Ευρωπαϊκού θεσμού, αφού εμεί δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την κακή πολιτική των κυβερνήσεων. Νομίζω λοιπόν ότι για μια ακόμη φορά είναι απαραίτητο να πούμε σε όλους ότι υπάρχει συνένεση στην οικονομική βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά ένα φορολογικό πολλαπλασιαστή. Αυτό το δείγμα είναι θετικό. Λίγες είναι οι εξαιρέσεις στη βιβλιογραφία. Η συνένεση λοιπόν Λέω ότι αν υπάρχει θετική ε, ενίσχυση υπάρχει ανάπτυξη. Αν υπάρχει περιορισμός μειώνεται η ανάπτυξη. Και λόγω αυτού του θετικού λοιπόν ε, φορολογικού πολλαπλασιαστή, διάφορε κυβερνήσει όπω τη είπα στη Γερμανία, στη Γαλλία, έχουν ληφθεί αποφάσει να, ε, να χρησιμοποιηθούν κάποιε πολιτικέ οι οποίε τελικά αύξησαν το έλλειμμα. Διότι ήξεραν ότι οι πολιτικέ αυτέ βοηθούσαν. Γιατί λοιπόν σε άλλε περιόδους όταν έχουμε δύσκολου καιρού, γιατί θα μπορούσε να βοηθήσει μια τέτοια πολιτική που έχουμε εδώ όπως είπατε τον κίνδυνο τη διπλή ύφεση. Γιατί υπάρχει αυτός ο γιατί εφαρμόζουμε όλοι τι λάθος πολιτικές. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν μπορούμε να έχουμε αυτόματισμού στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική πολιτική. Υπάρχουν καλές και κακές φορολογικέ πολιτικές και θα πρέπει να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητά του και μετά να τι κρίνουμε. As as Και θα πρέπει η εκτίμηση αυτή να γίνει το συντομότερο δυνατό. Δύο πράγματα πρέπει να πούμε. Το πρώτο, να θυμίσουμε ότι η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη και ότι η δημοκρατική διαδικασία έχει ε, οδηγήσει την έξω να προσπαθεί να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό. Το λέει η συνθήκη. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε η ΕΚΤ που είναι ουσιαστικά στην εφηβική ηλικία ακόμη, να ενηλικιωθεί. Και αν τη ζητείτε να συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις ή να συντονίζει το έργο των κυβερνήσεων, τότε όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Όλοι είμαστε ενήλικες, ανεξάρτητοι το δείχνουμε καθημερινά. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με την ΕΚΤ. Πρέπει όμω να γίνεται πάντοτε σεβαστή η ανεξαρτησία τη. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να αναφέρω είναι ότι δεν υπάρχει ε, ένα μέτρο για όλους ή μία πολιτική για όλους, άρα δεν υπάρχει ένας φορολογικός κανόνας που να ισχύει για όλους. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Γι' αυτό και εσείς θελήσατε να υιοθετήσετε αυτούς τους δείκτες μακροοικονομικών ανισορροπιών, έτσι ώστε να μπορούν να καταλάβουν και οι πολίτες ότι πρέπει να έχουμε διαφορετικές φορολογικές πολιτικές ανάλογα με την περίσταση. Ίσως δηλαδή σε μια συγκεκριμένη περίσταση να είναι καλή η πολιτική φορολογική, αλλά όχι σε μια άλλη περίσταση. Αλλά δεν υπάρχει μία και μόνο ε, πολιτική φορολογική που να είναι καλή για όλους. Τώρα, ποιε θα μπορούσαν να είναι οι μελλοντικέ βελτιώσει. Ελπίζω στο μέλλον να είμαστε σε θέση να δούμε κυβερνήσεις οι οποίες θα έχουν εμπιστοσύνη στην ΕΚΤ και ΕΚΤ να έχει εμπιστοσύνη βέβαια στις κυβερνήσεις, να υπάρχει συνεργασία χωρίς ε, συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ τους. Και αυτό που πρέπει να φροντίσουμε είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στο επίπεδο της ΕΚΤ, να δημοσιεύονται τα πρακτικά γιατί μπορεί και ο ιδιωτικό τομέα να θέλει ενημέρωση για το τι συζητείται στο επίπεδο τη έκτη, τι συμβαίνει. Δεν μα νοιάζει τι γίνεται με τη συνένεση. Η δημοκρατία σημαίνει διάλογο. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε. Την, ε, το διάλογο που διαμείβεται. Και μια τελευταία μεταρρύθμιση. Κάποιοι μιλάνε για τον χρυσό κανόνα τον δημόσιο οικονομικό, τον αυθεντικό κανόνα, όπου οι δημόσιε επενδύσεις μπορεί ίσως να χρηματοδοτηθούν μέσω των κρατικών ομολόγων. Εγώ νομίζω ότι είναι όριμος ο καιρός να το ξανασκεφτούμε. Γιατί να μην είναι αυτός ο χρυσό κανόνας για όλες τις επενδύσεις, αλλά να σκεφτούμε ποια είναι η καλή πολιτική, ποιο είναι το καλό φορολογικό σύστημα ή οι χρηστές δαπάνες. Αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον. Υπάρχουν ε, διάφορες αναγκαιότητες και επίγουσες καταστάσεις. Ε, πρέπει, παραδείγματος χάρη, να βελτιώσουμε τη σχέση μεταξύ ΕΚΤ και κυβερνήσεων. Και πρέπει να ξανασκεφτούμε τις ευρωπαϊκές μας πολιτικές για να μπορούμε να μετρήσουμε και την αποτελεσματικότητά τους. Ευχαριστώ. είναι οι ομιλητές Κλίντς, Ιντβελτ και Ούντο Μπόλτμαν. I've got Annie, Liam, um, Werner, Mr. Dorfman. Anybody else? So the list is Wolf, Sophie, Udo K, Annie, Liam, Werner. Λοιπόν, η λίστα ξεκινάει με τον κύριο Γούλφ. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να σας ενώσω σε ενότητες, διότι έχουμε μόνο 35 λεπτά, οπότε θα πάρω τρεις ενότητες. Πρώτα ο Βόλφ. Ευχαριστώ. Καταρχήν μερικά σχόλια στον Γάλλο καλεσμένος μας. Αυτό που είπατε μου θυμίζει την πρόταση ότι αν κάποιος έχει φοβερό πονοκέφαλο γιατί πιε πολύ κρασί, πιες νερό και θα στρώσεις. Δεν αντιλαμβάνουμε δηλαδή να είναι πολύ λογικό το σχόλιο σας αυτό. Μετά όσον αφορά την ανεξαρτησία της ε, ΕΚΤ. Αντιλαμβάνομαι ότι είστε υπέρ της ανεξαρτησίας, αλλά βλέπουμε ότι με ε, την συνεργασία τουλάχιστον ε, στο, στα μάτια πολλών η ΕΚΤ έχει χάσει ένα μέρος της ανεξαρτησίας της. Οπότε εφόσον μπορείτε να συνεργάζεστε και να μην αμφισβητείτε ε, ε, δεν είναι δυνατόν να συνεργάσετε και να μην αμφισβητηθεί η ανεξαρτησία σας. Προς τον κύριο Στάρκ. Νομίζω ότι πολύ σωστά Είχατε ορισμένες αμφιβολίες για το εάν αυτή η νέα οικονομική διακυβέρνηση και το six-pack θα λειτουργήσουν σωστά στην πρακτική. Είναι εξαίσιο στη θεωρία, αλλά να δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Και εγώ έχω μεγάλες επιφυλάξεις, διότι οι αρχηγοί κρατών μέχρι στιγμής δεν έχουν θελήσει να ακολουθήσουν την κοινοτική προσέγγιση, βασίζονται σε διακυβερνητικές μεθόδους και ε, πρέπει να ε, έχουν την τελευταία λέξη. Ε, δεν θέλουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεμβαίνει και να κινείται αποφασιστικά. Τι θα γίνει όμως αν την επόμενη φορά δούμε αυτό που διαπιστώσαμε και την πρώτη φορά, ότι υπάρχει μία, ότι δεν σε τα συμπεφωνημένα οι ε, άλλοι, δεν υπάρχει αντίδραση, υπάρχει ένα δεύτερο ε, πλάνο, ένα πλάν B, διότι αυτό το ότι η Ευρώπη είναι πολύ σημαντική, δεν μπορούμε να τη διακινδυνεύσουμε κάνοντας αυτό και εκείνο, δεν με ικανοποιεί. Ε, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που περιμένω και προσδοκώ. Και τέλος, πώς αξιολογείτε τον ε, κίνδυνο της ε, ε, περαιτέρω ενώσεως στην Ευρωζώνη διότι μπορεί να σπάσουμε την, Ευρωζώνη στα δύο, την Ευρώπη στα δύο αυτούς που είναι στην Ευρωζώνη και αυτούς που δεν είναι η κυρία Ίντβελτ Συμφωνώ με τον Βολφ και τον κύριο Στέρκ γιατί με, με εξέπληξε η εισήγησή σας, η εισήγηση του κυρίου Κρέλ, διότι μπορούμε να έχουμε όσα σύμφωνα και συμφωνίες θέλουμε. Εάν δεν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή και αν δεν υπάρχει πολιτική θέληση για την εφαρμογή τους, όπως είπε και ο Βόλφ, τότε δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, όπως έχει και ο τίτλος της παρουσίασής σας. Και η διαχείριση μέσω ομοφωνίας είναι αδύνατη. Φτάσαμε στα όρια μας. Και μου κάνει εντύπωση το ότι λέτε ότι πρέπει να έχουμε ένα από τα ίδια. Είπατε επίσης ότι δεν υπάρχουν ενιαίες λύσεις για όλα. Αν όμως δείτε το δολάριο, βλέπετε ότι και η ΕΠΑ δεν είναι μια ομοιογενής ε, περιφέρεια, όμως έχουν μία κυβέρνηση και αυτό εμπνέει εμπιστοσύνη. Γιατί δεν υπάρχουν ε, βέτο από τα διάφορα κράτη γι' αυτό μπορούν να αποφασίσουν, έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν κάτι που εμείς ε, δεν έχουμε. Έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Στάρκ. Είπατε ότι θα πρέπει να απαρνηθούμε τα ευρωομόλογα, μα είναι και θέμα χρονισμού, γιατί αν δημιουργήσουμε ένα νέο πρότυπο, μία νέα πρότυπη ευρωζώνη που θα είναι περισσότερο ομοσπονδιακού χαρακτήρα, τότε τα ευρωομόλογα δεν θα είναι ένα μέσον προς αυτή την κατεύθυνση. Και υπάρχουν και προτάσεις οι οποίες ε, επιπλέουν και υφίστανται σε σχέση με τη μείωση των κινδύνων από τα ευρωομόλογα. Δεν θεωρείται όμως ότι θα ήταν αναπόσπαστο μέρος αυτού του συστήματος ο Ούντο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την πρώτη δήλωση του Βολφ Κλίντς, ο οποίος ε, είχε αναφερθεί εις ε, τις προβλέψεις της Commerzbank και έχω την εντύπωση κύριε Στάρκ ε, ότι το πόσο θα προχωρήσει η Ευρωζώνη του χρόνου θα έχει λιγότερη σχέση με την κατανάλωση νοπνευματοδών αλλά ότι μπορεί να βρεθούμε σε μία βαθιά ύφεση και ε, γι' αυτό έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Στάρκ και τον κύριο Κρέλ σχετικά με την ε, ανακοίνωση των υπουργών του G20 το περασμένο Σαββατοκύριακο όπου είπαν τι θα έπρεπε να κάνουν ε, οι οικονομίες και αναφέρω ένα σχόλιο ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές για να μετακινηθούν προς ανάπτυξη που βασίζεται στην εσωτερική ζήτηση και στην αποταμίευση. Θα ήθελα λοιπόν οι δύο κύριοι να μου πούν ε, πώς αξιολογούν τα σχόλια αυτά. Δηλαδή πρέπει να δημιουργηθούν πλεονάσματα, συμφωνείτε με τη μέθοδο αυτή και πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτά τα πλεονάσματα. Και επίσης όσον αφορά αυτούς ε, οι οποίοι ε, μπαίνουν στην κρίση, δηλαδή τα κράτη της Νοτιού Ευρώπης και Ευρωζώνης ε, τι πρέπει να γίνει γιατί αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Στάρκ. Ιδίω διότι ε, το θέμα αυτό ε, επέμεινε ότι έπρεπε να το συζητήσουμε και η ερώτησή μου εδώ αναφέρεται στην ακραία κατάσταση. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή για να προστατεύσουμε την Ευρωζώνη. Μας λέτε ότι δεν πρέπει να επέμβει η έκτα, ε, ε, ε, όχι ευρωμόλαγα Τι θα κάνουμε, θα αφήσουμε να καταρρεύσει η Ευρωζώνη, αυτή είναι η εναλλακτική λύση. Κάπως θα πρέπει να το σκεφτούμε, θα ήθελα να ξέρω πώς διαβλέπετε το νέο θεσμικό πλαίσιο, πού τοποθετείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πόσο ε, θα βρίσκεται ε, σε σχέση με το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα προγράμματα τα οποία σκέφτεστε. Πολλές ερωτήσεις υποβλήθηκαν, αλλά προβλέπετε και δεύτερος γύρος. Ε, δεν έχετε πολύ καιρό για να απαντήσετε. Ο Γιούργεν μπορεί να αρχίσει σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Κλίντς. Κατά πόσο η οικονομική διακυβέρνηση μπορεί να εφαρμοστεί και τι θα συμβεί εάν οι κανόνες δεν εφαρμοστούν. Είπα σαφώς στην εισήγησή μου ότι αυτό που έχουμε επιτάπιος δεν είναι αυτό που ζητήσαμε, που ζητήθηκε από την ΕΚΤ. Χρειαζόμαστε σαφέστερους κανόνες και πιο σκληρούς για να επιληθεί η τρέχουσα κατάσταση και για να προωθήσουμε και την οικονομική διακυβέρνηση. Άρα υπάρχει το θέμα της εφαρμογής. Ε, τη στιγμή που υπάρχει μία κατάσταση de facto, έχουμε πρόβλημα. Η εφαρμογή είναι ύψης της σημασίας και φτάσαμε στα όρια της ε, ομοφωνίας. Δεν θεωρώ ότι οι ΙΠΑ οι οποίοι έχουν ένα διαφορετικό πλαίσιο, έχουν άλλες δυνατότητες απόφασης, ζουν σε ένα ε, άλλο θεσμικό πλαίσιο και έχουν και εκείνοι προβλήματα έγκρισης. Όπως είδαμε και από την πράξη και από τις τελευταίες νομοθετικές πράξεις. Σε πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια. Αλλά χρειάζεται πολιτική θέληση για να εφαρμοστούν οι κανόνες και να, να εφαρμοστούν τα συμπεφωνημένα. Και με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το ρόλο που διαθέτει, θα μπορέσει να συνεισφέρει. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στην Επιτροπή και το Συμβούλιο τα ε, δικαιώματα και τα καθήκοντά τους. Θα πρέπει να μας γίνουν όλα αυτά μάθημα. Ως προς τα ευρωμόλογα, δεν αναφέρθηκα στους όρους υπό τις οποίους τα ευρωμόλογα είναι ένα ενδιαφέρον μέσο ή μηχανισμός. Διότι επί της ουσίας τα ευρωμόλογα αφορούν μία άλλη ε, διάρθρωση διακυβέρνησης και μέσα στα πλαίσια αυτής της σύγκλησης ή της ολοκλήρωσης τα ευρωομόλογα είναι ένα εφικτό μέσον, αλλά χρειάζονται διαφορετικές προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρξει μεταφορά εθνικής κυριαρχίας η οποία να ανατεθεί σε έναν υπερεθνικό, σε υπερεθνικό επίπεδο. Ως προς το ερώτημα του κυρίου Πούλμαν, σε επίπεδο G20, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν οι πλεονασματικές χώρες και τι ελληματικές, αυτό μου θυμίζει και εδώ εκφράζω την προσωπική μου άποψη, την κατάσταση το 78 στο, στους G7 στη Βόνη, όπου Μιλήσαμε για συγκεκριμένα θέματα ως προς ε, συγκεκριμένες χώρες, κάτι το οποίο δεν λειτουργήσε. Ε, ίσως λειτουργήσει σε επίπεδο G20, αλλά θα πρέπει να εναρμονιστούμε. Και το μεγάλο πρόβλημα αφορά τις ε, ελληματικές χώρες, όχι τις πλεονασματικές. Και δεν συμφωνώ με αυτή την ε, συμμετρία προσαρμογής που αναφέρεται αυτής. Χρειαζόμαστε μία ασύμετρη προσέγγιση, διότι τα βασικά προβλήματα αφορούν τις ελληματικές χώρες και θα πρέπει να τις εντομετωπίσουν αυτές οι χώρες ως προς την περιφέρεια και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν μιλάμε μόνο για φορολογική ολοκλήρωση. Θα ήταν πολύ απλουστευτικό να πούμε ότι η φορολογική ολοκλήρωση θα οδηγήσει σε συρρήκνωση της οικονομίας. Ακόμα και 70 χρόνια μετά τον Keynes δεν υπάρχει συμφωνία στους οικονομολόγους για το ρόλο του φορολογικού πολλαπλασιαστή. 70 χρόνια μετά τον Keynes και το τονίζω αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι η φορολογική και η διαρθρωτική, η δομική μεταρρύθμιση. Και επίσης μεγάλη σημασία έχει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης, η οποία θα πρέπει να αρχίσει. Θα πρέπει να πάρουμε αυτά τα στοιχεία, δηλαδή φορολογική ολοκλήρωση γιατί δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος. Οι αγορές ε, αντιδρούν διαφορετικά από ό,τι αντιδρούσαν μέχρι τα μέσα της ε, προηγούμενης διετίας. Και η ανοχή στο χρέος έχει μειωθεί, άρα οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν δέχονται ένα όλο ένα και διονγκούμενο χρέος και έλλειμμα. Αυτό δηλαδή που ζήσαν στο παρελθόν οι αναδιόμενες χώρες, το ζουν τώρα οι μεγάλες οικονομίες, το λεγόμενο start and stop. Οι αγορές λοιπόν δεν δέχονται αυτή την προσέγγιση πλέον. Δηλαδή δεν δέχονται αυτό το διονγκούμενο χρέος. Άρα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συνυπάρξουν και να συνάδουν σχετικά με τον μηχανισμό σε έξαρση. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή, όχι, όχι μακροπρόθεσμα τώρα, χωρίς ΕΚΤ ε, με EFSF και ESM. Ε, Απαντώ γερμανικά λέει ο κύριος Στάρκ. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να απαντήσουμε θετικά ότι η Ελλάδα θα πάρει την επόμενη δόση και αυτό είναι πολύ οξύ για να μπορέσει να υπάρχει βιωσιμότητα των χρεών στα πλαίσια του προγράμματος αυτού. Βέβαια, σχετικά με το EFSF, με την ευελιξία για τη μόχλευση, για τις ασφαλίσεις. Το EFSF δεν θα απαντηθεί από την ΕΚΤΑ, αλλά από τους πολιτικούς. Μετά, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για να μπορέσει να υπάρχει η δυνατότητα να θωρακιστούν εάν ενταθεί η κρίση. Αυτές είναι οι λύσεις τις οποίες εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Φοβούμαι ότι η παρουσίασή μου ήταν χειρότερη από το γραπτό κείμενο. Μήπως καλύτερα να διαβάσετε το γραπτό κείμενο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν μου άρεσε αυτό το επιχείρημα με το αλκοόλ και το πονοκέφαλο, γιατί ε, πρέπει να αναρωτηθείτε γιατί κάποιος είναι αλκοολικός. Δηλαδή γιατί σήμερα τόσες πολλές χώρες έχουν τόσο υψηλά ελλείμματα. 17 χώρες στην Ευρωζώνη. Μία μόνο έχει συμπεριφερθεί άσχημα επί σειρά ετών η Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να ελέγξουν τα δημόσια οικονομικά τους, αλλά θα έπρεπε να τους έλεγχαν ήδη από το 2002. Πρέπει αυτό να αλλάξει τώρα. Εντάξει. Υπάρχουν όμως άλλες 16 χώρες. Πριν την ε, κρίση, πριν από τέσσερα χρόνια, σε καμία περίπτωση ε, δεν είχε περάσει κάποια χώρα το 3%. Ήταν καλά τα δημόσια οικονομικά με βάση τους τότε κανόνες. Ίσως να μην ήταν σωστοί κανόνες, αλλά τηρούσαν τους κανόνες οι χώρες. Άρα έγιναν αλκοολικές εντό αγωγικών, επειδή υπήρξε αυτή η παγκόσμια κρίση. Και σήμερα δεν σκεφτόμαστε να χρησιμοποιήσουμε νέα φορολογική όθηση, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ ε, άρρωστη η χώρα από τον αλκοολισμό. Και δεν έχουμε μόνο το δημόσιο ε, χρέος. Έχουμε και το ιδιωτικό. Και υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και τον είπα για παράδειγμα. Δεν είχαν αυτό το χρέος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως υπάρχουν αυτά τα περιθώρια έλλειμμα Καταλαβαίνω ότι οι αγορές είναι αυτές οι οποίες μας λένε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε υψηλό έλλειμμα ή υψηλό χρέος. Ενώ ταυτόχρονα ζητούν ανάπτυξη. Φυσικά δεν μπορώ να σας πω ότι αύριο θα έχουμε ανάπτυξη, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι διαφωνώ πλήρως με τον καθηγητή Στάρκ. Αλλά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ε, συνένεση για αυτό το θετικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, στη βιβλιογραφία τόσα ε, διατριβές και τόσα συγγράμματα, το ίδιο πράγμα λένε ουσιαστικά, ότι είναι θετικό, υψηλό μεν αλλά θετικό. Και πραγματικά και από τον ΩΣΑ και από το Διεθνές Ταμείο υπάρχουν συγγράμματα So, did, did they... Yes, but I'm sorry, but I think... Δυστυχώς δεν ακούσαμε το ερώτημα. Τέλος πάντων, γιατί είμαστε αλκοολικοί. Αυτό είναι το ερώτημα. Είχαμε μια κρίση και έπεται και επόμενη. Τι θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Δηλαδή απελπισία, έλλειψη εμπιστοσύνη ε, στους θεσμούς. Πώς θα εξηγήσουμε τότε στους πολίτες μας ότι χρησιμοποιήσαμε πριν από δύο-τρία χρόνια φορολογικές πολιτικές και παρά ε, τις συνθήκες και το ότι είναι ε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχω απαντήσεις να δώσω, απλά ερωτήματα θέτω σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεργασία. Εγώ έλεγα, σε σχέση και με αυτό που είπατε, κάπως εξαναγκάστηκε να συμμετέχει η έκτα σε κάτι που ίσως δεν ήθελε. Ίσως δεν ήθελε να συμμετέχει η έκτα. Αν η αρχική κρατών και κυβερνήσεων ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με του πολίτε με το λαό, πούν ότι ναι, ξέρουμε ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι ανεξάρτητη, ε, φόρ ζωή. Θα πρέπει να παρακολουθεί τη σταθερότητα των τιμών, γιατί το λέει το καταστατικό τη η εντολή τη. Ίσως τότε η ΕΚΤ δεν θα σκεφτόταν ότι αν ζητήσουμε τη διαπραγμάτευση, τη συνεργασία με άλλου θα σκεφτούν ότι τη βάζουμε να κάνει κάτι που δεν θέλει. Με βάση τον ΝΑΣ, που πάντοτε αυτό που προτείνει είναι ε, μια κατάσταση στην οποία κερδίζουν όλοι, αυτό λέω εγώ. Μια κυβέρνηση προσπαθεί να συζητήσει με την ΕΚΤ και ακούμε ότι η ΕΚΤ δεν είναι ανεξάρτητη ή θα μπορούσε να μην είναι ή ε, αντιμετωπίστε σαν να μην είναι. Όχι, έχουμε ένα σχέδιο, έχουμε ένα project και αυτό το σχέδιο είναι το ευρώ. Πρέπει λοιπόν να επαναλάβουμε ότι χρειάζεται η ΕΚΤ, γιατί ε, στην παγκόσμια κρίση τα κατάφερε περίφημα, αλλά πρέπει να είναι ανεξάρτητη, πρέπει να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός. Και αν φτάσει ε, να έχουμε σταθερότητα των τιμών, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Ε, δεν ξέρω τι κάνει η ΕΚΤ, εγώ είμαι αισιόδοξο. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε σε ό,τι αφορά το είναι επιβολή, το enforcement, δεν έλεγα ότι δεν... Ε, ουσιαστικά δεν ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Απλά έλεγα ότι μεταξύ όλων αυτών τα οποία θα πρέπει να παρακολουθούνται, ίσως θα πρέπει να διερωτηθούμε γιατί εφαρμόζουμε φορολογικές πολιτικές. Ίσως έχει δίκιο ο καθηγητής Στάρκ. Ίσως είναι αρνητικό ο ε, φορολογικός πολλαπλασιαστής. Άρα πετάμε στα σκουπίδια ε, τη φορολογική πολιτική, δεν χρειαζόμαστε φόρους, δεν χρειαζόμαστε δαπάνες. Αφού είναι αναποτελεσματικό, ας το σταματήσουμε. Γιατί το χρησιμοποιούμε, γιατί χρησιμοποιούμε αυτές τις πολιτικές. Μια ερώτηση είναι αυτή. Και σε ό,τι αφορά το έλλειμμα και το πλεόνασμα τώρα. Αυτή είναι η συμμετρία που έχει να κάνει με, αυτή, με τον πίνακα επιδόσων, το scoreboard επαρκείς ή ανεπαρκείς αποταμιεύσεις ή εξοικονομήσεις. Μια χώρα που είναι σε κρίση μειώνει ε, το έλλειμμα. Ε, είναι μια επιλογή. Αν υπάρχει μια ε, από έξω. Και νομίζω ότι αυτό προτείνει και η ομάδα των 20, το G20 ο πρόεδρος. Λοιπόν, θα πρότεινα οι πέντε ομιλητές που απομένουν να κάνουν τις ερωτήσεις τους μαζί και αν είναι τυχεροί μπορεί και να ακούσουν και τις απαντήσεις, αρκεί να μακρηγορήσουν. Και οι Άννη, Βέρνερ, Λίαμ και Χέρμπερτ είναι οι πέντε ομιλητές. Ο Βέρνερ πήγε πιο πάνω στη λίστα γιατί δεν είχε μιλήσει κάποιο άλλος από το ΕΛΚ. Okay. Είπα ότι είχαμε, θα είχαμε εδώ τους ε, πάνελ, τα μέλη του πάνελ και νομίζω ότι ε, όλοι μου ε, είπαν να υποβάλω ένα ερώτημα σε εσά, κύριε Στέρκ. Πώς ένα αξιότιμο μέλος της ΕΚΤ στην ουσία αποχώρησε από την ΕΚΤ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους αποχωρήσατε. Ιάννη. Σάρον, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, τα μέλη του πάνελ. Έχουμε διάφορα επίπεδα συζήτησης και έχουμε πολλά να μάθουμε από την τρέχουσα κρίση για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα έχει η νέα οικονομική αρχιτεκτονική. Αλλά ως προς τη διαχείριση της κρίσης, αν δεν την διαχειριστούμε σωστά και συνεκτικά, καθώς και με συνέπεια, όλες αυτές οι συζητήσεις και τα μέτρα σε σχέση με τη νέα οικονομική διακυβέρνηση θα είναι χωρίς σημασία και περιεχόμενο. Θα ήθελα να ρωτήσω όλα τα μέλη του πάνελ το εξής. Τρεις μήνες πριν είχαμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θεωρήθηκαν ιστορικές για την διαχείριση, για την ε, μη παράταση και διάδοση της μόλυνσης και απάντηση στο ελληνικό ζήτημα. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε έναν νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πάλι θα θεωρηθεί ιστορική σημασίας. Απλή ερώτηση. Τι δεν πήγε καλά μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου και τι θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε το επικείμενο Συμβούλιο να είναι πραγματικά επιτυχές και να μπορέσει να διαχειριστεί τελειωτικά την ε, κρίση. Ως προς τη φερεγγιότητα ή μη της Ελλάδας γίνονται πολλές συζητήσεις για την ε, αναδιάρθρωση του χρέους και σε σχέση με το PSI θα ήθελα τις απόψεις σας. Θεωρείτε ότι η αποφάση της 21ης Ιουλίου για το PSI ήταν επαρκής ή πιστεύετε ότι μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης λύσης αυτό το σκέλος θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης. Ε, Ευχαριστώ. Έχω πολλές ε, ερωτήσεις. Ε, καταρχήν δεν με έπεισε η επιχειρηματολογία του κυρίου κρέλ ότι το να έχει κανείς χρέη δεν είναι λύση και μας το έχει αποδείξει και η οικονομική ιστορία. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε και το Σύμφωνο Σταθερότητος με τους τότε αριθμούς. Ήταν ε, η κατάσταση όταν δημιουργήθηκε το Σύμφωνο Απασχόλησης και Σταθερότητος με τα ποσοστά αυξήσεως της προηγουμένης δεκαετίας 3% και τώρα το ποσοστό θα πρέπει να είναι χαμηλότερο και όχι ψηλότερο ως προς τη δημιουργία χρεών. Ε, μία άλλη παρατήρηση σχετικά με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, είμαι εισηγητής για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, αλλά ε, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Προέδρου της 21ης Ιουλίου του 2010, ο οποίος γυρίζει το ο ρολόι πίσω χωρίς να έχει επιλεγεί ε, νέο κογκρέσο δεν ε, ξέρω πού θα πάμε. Μ' αρέσουν οι ιδέες που παρουσιάσατε αλλά βλέπω ότι υπάρχει μία έξαρση των εθνικών εγωισμών τα τελευταία χρόνια και η ψηφιακή μέθοδος ε, που δεν είναι λόγο δεν προσανατολίζεται προς την κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κατά τη γνώμη μου δεν είναι σε θέση να παράσχει ε, τις οργανωτικές προϋποθέσεις ούτε την Ελλάδα ήλεγξε ούτε κανέναν άλλον υπάρχουν πολλές παραλήψεις καμία διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και δεν μιλάμε μόνο για τα κράτη-μέλη εδώ αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κύριε Στάρκ σχετικά με την ε, ε, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών οι Αμερικανοί μόλις μόλις ολοκλήρωσαν αυτή τη διαδικασία αλλά οι Ευρωπαίοι ακολούθησαν άλλη οδό. Θεωρείται ότι το αμερικανικό σύστημα ήταν πιο επιτυχές και ε, μία ε, εθελοντική ε, έξοδος από την Ευρωζώνη θα μπορούσε να συζητηθεί αν η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της. Με συγχωρείτε αγαπητοί συναδελφοί αλλά δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν απαντήσεις αν δεν είστε πάρα πολύ πολύ σύντομη. Έχω δύο ερωτήσεις. Κύριε Κρίλ, αυτή η συζήτηση για τους πολλαπλασιαστές είναι πολύ σημαντική. Αν θεωρήσουμε ότι θα υπερισχύσει η αρχή του πολλαπλασιαστή και νομίζω ότι υπερισχύει σε σχέση με την ε, ε, εξίσωση, την λεγόμενη εξίσωση Ρικαρδιέν. Αυτό σημαίνει συρίκνωση των ε, δαπανών και αυτό οδηγεί σε ύφεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί. Στη Γαλλία για το 2012 μιλάμε ότι περνάμε από το 2,25 σε 1,75 και οι μακροοικονομολόγοι θεωρούν ότι το 2012 θα είμαστε στο 0,8%. Αυτό σημαίνει ότι υπολοιπόμαστε κατά 10 δις εσόδων. Εάν λάβουμε υπόψη και την αύξηση φόρων που θα γίνουν του χρόνου, διότι αναθεωρήσαμε το δίκτυο ανάπτυξης για να φτάσουμε στο κριτήριο του 4,6% του δημοσίου ελλείμματος και 3% ε, αντίστοιχα 12 και 13 θα είναι πολύ δύσκολο. Ποιο θα, ή ποιο θα ήταν το στοιχείο για να έχουμε μία συρρήγνωση κατά 20 δις εάν η γαλλική κυβέρνηση αρκεστεί στο κριτήριο του 3% του, το 2013 και προς τον κύριο Στάρκ από πλευράς ε, ΕΚΤ που δεν αποφασίζει για τη δημοσιονομική πολιτική το βραβείο Νόμπελ μας είπε ότι μια χώρα σαν τη ΣΥΠΑ δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Εσείς ζητήσατε από τα κράτη να απαρνηθούν αυτή την εθνική κυριαρχία του, την οικονομική εθνική κυριαρχία του. Πιστεύετε λοιπόν ότι η εθνική κυριαρχία είναι χρήσιμη ή όχι. Θα ζητήσω από τα μέλη του πάνελ να απαντήσουν σε ένα λεπτό και τα υπόλοιπα θα μας τα αποστείλουν γραπτός. Εγώ έχω μία πολύ σύντομη ερώτηση στον καθηγητή Στάρκ. Είπατε ότι στην εφαρμογή της μακροοικονομικής ε, εποπτείας ε, διαβλέπεται προβλήματα και ε, αντιλαμβάνομαι ότι με την νέα νομοθεσία θα πρέπει αυτά τα θέματα να ρυθμιστούν. Πιστεύετε ότι αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί είναι αποτελεσματικά ή ότι η, βάση, η νομική βάση που χρησιμοποιούμε δεν είναι η ενδεδειγμένη. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο πρώτο στον κύριο Στάρκ γιατί έχουν δοθεί ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και είμαι βέβαιη ότι όλοι θέλετε να ακούσετε τις απαντήσεις και ε, γι' αυτό ένα λεπτό θα έχει ο καθένας. Δέκα δευτερόλεπτα για το θέμα που συζήτησε και στον πρώτο γύρο, η ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Η ανεξαρτησία της ΕΚΤ ποτέ δεν έχει αφισβητηθεί. Πρώτον. Δεύτερον, το να ζητώμε να κάνει περισσότερο η ΕΚΤ θα, ε, είναι, ε, ε, θα θέσει κίνδυνο την ανεξαρτησία της. Δεύτερον, ότι ανακοινώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου από την ΕΚΤ ότι θα αποσυρθώ όταν ε, θα βρεθεί ο αντικαταστάσης μου είναι για ε, προσωπικούς λόγους. Είμαι στο, στη θέση μου και θα παραμείνω μέχρι το τέλος του χρόνου και ε, πολύ πιθανόν στο τέλος του χρόνου θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Αλλά προς το παρόν εδώ βρίσκομαι και δεν νομίζω ότι αξίζει να γίνονται συζητήσεις τι έγινε μεταξύ του Ιουλίου και του Οκτωβρίου. Έλλειψη εφαρμογής. Χρειάστηκε πολλή χρόνος να εφαρμοστούν αυτά τα οποία απεφασίστηκαν στις 21 Ιουλίου και αυτό δημιούργησε ένα κλίμα μεγάλης ασταθείας και αβεβαιότητος και αυτό είναι το σημείο κλειδί. Όσον αφορά την Ελλάδα τι αποφασίστηκε στις 21 Ιουλίου για την Ελλάδα 21% περικοπή το οποίο δεν εφαρμόστηκε όλες οι εργασίες έπρεπε να έχουν επιταχυνθεί για να υπάρχει μια γρήγορη λύση όταν θα είναι η κατάλληλη στιγμή σχετικά με την ερώτηση του κυρίου Λάνιεν πολύ σωστά υπάρχει αποτελεσματικότητα και στο εθνικό και στο υπερεθνικό επίπεδο Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα σε μία πολύ σοβαρή κρίση του κυριάρχου κρέους αλλά αυτό οφείλεται διότι στις καλές εποχές δεν εφαρμόστηκαν πλήρως οι κανόνες και όταν οι κυβερνήσεις δεν σεβάστηκαν τις υποχρεώσεις τους και υπερέβησαν τους στόχους σας και οι διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, δεν χρησιμοποιήθηκαν οδηγηθήκαμε εκεί. Μετά ε, σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είναι ε, κάτι το οποίο στην Αμερική επέτρεψε μεγαλύτερη αξιοπιστία. Τώρα έχουμε κάνει δύο στρες τεστ στην Ευρώπη και το θέμα είναι ακόμη ε, να εξελίξει. Δηλαδή οι αγορές δεν θεωρούν ότι έχουν επιτύχει. Ε, παρακαλώ συντομεύστε λέει η πρόεδρος. Ναι. Ε, θα υπήρχαν ανεξέλεγκτες επιπτώσεις αν η Ελλάδα εγκαταλείψει την Ευρωζώνη και τέλος σχετικά με το μακρο ε, οικονομικό βαθμολόγιο, το scoreboard, θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευελιξία. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο σε λίγους δείκτες. Τεχνικά ε, η συνεδρίαση έχει τελειώσει και γι' αυτό τώρα θα ζητήσω από τον κύριο να απαντήσει πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι οι αυτόματες ε, κυρώσεις είναι συζητήσιμες αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αλληλεγγύη δεν θα πρέπει να είναι αυτόματη, θα πρέπει να γίνει αυτοματοποιημένη, να αυτοματοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν άμεσα οι αποφάσεις, ιδιαίτερα για το ελληνικό θέμα. Τώρα, κατά πόσο... This Κατά πόσο θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ψηλότερο χρέος και κατά πόσο θα ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι υπάρχουν καταστάσεις όπου θα ήμασταν καλύτερα με, με πολύ χαμηλότερο χρέος, αλλά θα πρέπει να δούμε τους συσχετισμούς. Ως προς το ερώτημα του Γάλλου συναδέλφου, δεν ξέρω για τον πολλαπλασιαστικό δίκτυο Πώ ε, πώς ισχύει στη Γερμανία, αλλά είναι 0,8 μέχρι 1,8. Βράχει πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ε, ο Αντρέι Ρικάρτο θέλει κάτι να πει. Τι δεν πήγε καλά λέει ο κύριος Καμπράλα. Νομίζω ότι υπήρχε κακή κατανομή κεφαλαίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέβαλε την ε, αναγνώριση αυτών των ε, ζημιών. Ως προς την ε, νέα κεφαλαιοποίηση των τραπεζών νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μέσα στα πλαίσια της εξηγίασης των τραπεζών. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ζήτησα από το, τα μέλη του πάνελ να επεκταθούν γραπτός, αν το επιθυμούν, γιατί δεν είχαμε χρόνο και οτιδήποτε λάβουμε θα σας το διανύμουμε βεβαίως. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις προς το τέλος όταν δεν υπάρχει χρόνος για απαντήσεις. Αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτές κατά τη γραπτή διαδικασία. Τώρα έχουμε συνεδρίαση συντονιστών Γι' αυτό όσοι δεν ε, πρέπει να παρεπρεθούν θα ήθελα να αποχωρήσουν σύντομα. Ευχαριστώ.